Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7. Bericht Brandner. Πάμε στο σημείο αυτής της μέσης διάταξης. Έχουμε δύο εκθέσεις Μπράτνερ. Ε, λίγες είναι κιόλας, λέει ο πρόεδρος. So, zuerst reden wir Ωραία, λοιπόν, πρώτα συζητάμε την ε, οδηγία 2409 για την εναρμόνιση των προποθέσεων διαφάνεια αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότε των οποίων οι κινητέ αξίε έχουν εισαχθεί προ διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά καθώ και τι οδηγίε και τι οδηγίε 2007-14 τη Επιτροπή. Ο εισηγητή έχει τίποτα να μα πει, ή η εισηγήτρια. Όχι, ψηφίζουμε λοιπόν. Antrag 8. Wer ist dafür? Παριθμόν 8 υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεν με προσέχετε, δεν με προσέχετε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 19 υπέρ 25 κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 3 ε, έχει αποσυρθεί στη συμβαστική 2 υπέρ κατά απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία. 9. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται επίση. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται με την ίδια 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική υπαριθμόν 1. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Υπαριθμόν 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 2 έχει αποσυρθεί. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για το σχέδιο στο σύνολό του. mit 22 zu 25 abgelehnt. 22 υπέρ, 25 κατά, απορρίπτεται. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια πράγμα πάλι ποτέ, αλλά κάθε τι, κάποτε. Έχει μια αρχή. Πάμε τώρα. Τι θέλετε. 25 κατά 22 υπέρ ήταν η ψήφος. Δεύτερη έκθεση τώρα. Τι πάλι της κυρίας Βρόντσινας. Βλέπω από τη δική μου τουλάχιστον ομάδα κάποια θετικά πρόσημα, αλλά θα δούμε. Κυρία Μπρόντσινας. για, το, για την πρώτη τροπολογία που έχουμε στην σειρά των ε, ψηφοφοριών. Δεν έχω βάλει πρόσημο γιατί είναι εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας. Και γι' αυτό ουσιαστικά θα πρότεινα να μην ψηφιστεί καν. Αλλά μπορείτε να τη θέσετε στη ψηφοφορία αν, θεωρείτε, το θεωρείτε σκόπιμο. Πάντως είναι θέματα της νομικής επιτροπής, δεν είναι της δικής μας. Καλώς, λοιπόν, θέλετε να μας εξηγήσετε το γιατί. Ναι, είναι πολύ ευρύ το πεδίο της ε, οδηγίας. Μιλάει για θέματα επιχειρήσεων και άλλες λεπτομέρειες, τις οποίες ε, δεν έχουμε εμείς καμία σχέση δουλειά μας, ούτε και η Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων. Δεν έχει θέση εδώ στην Επιτροπή, την ΑΦΕΤ. Anyone else to say something about it? Frau Karens? Θέλει κανείς να λάβει το λόγο, κυρία Κάρενς είναι εδώ. Herr Karens. Yeah. Karens Herr Karens. Κύριος Κάρενς, παρακαλώ. Yeah, Please could you explain your position to that? Uh, thank you, Mr. President. I think uh, this point is beyond debate. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι για αυτή τη συζήτηση πάντως, Πρόεδρε. Είχαμε πει στο προσχέδιο ότι ήταν και αυτό πέραν αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Δηλαδή έχουμε την ίδια λογική. Νομίζω ότι είναι αργά να κάνουμε τέτοια σχόλια και θα πρέπει να προχωρήσουμε την ψηφοφορία. Καλώς ψηφίζουμε. Την 30. Υπέρ. Υπέρ της 30. Κατά. Ας απολυθεύσουμε. Υπέρ, λέει ο πρόεδρος. Πέρας. 36 υπέρ 9 κατά. Η 31 έχει αποσυρθεί, συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Πέρας. 23 υπέρ, 27 κατά. Στην 4 υπέρ. Κατά. Με την ίδια προψία απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39-40 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ. Α, όχι αυτή. 41 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται νομίζω. Επαληθεύουμε. Πέρα στις προφορίες. Απορρίπτεται. Με την ίδια πλειοψηφία. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές το. 44 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Πέρας. 27 υπέρ, 23 κατά. 45 τώρα, όχι καταπίπτει. 7 και 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 47 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 48 καταπίπτει. 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 50 καταπίπτει. Η 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Πέρασε φορές. 27 υπέρ, 24 κατά. Εγκρίνεται. 9 και 53 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 10 και 54 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 12 και 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 13 και 57 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 14 και 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 έχει αποσυρθεί 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 και 61 υπέρ κατά απορρίπτεται 62 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 17 και 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές επαληθεύουμε. Πέρασε προφορία. 21 υπέρ, 29 κατά η ψήφη, απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 και 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ Συγγνώμη, υπέρ, λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 λέει ο πρόεδρος. Υπέρ, κατά αποχές. Ο πρόεδρος συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Υπαριθμόν 1 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά. Επαληθεύουμε την 24. 24 λοιπόν. Ε, και την 1, εντάξει. Την 1 πρώτα. Τροπολογία 1 ελέγχουμε. Πέρας. Απόρριπτεται. 26 υπέρ, 27 κατά. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και έτσι περνάμε στην υπαριθμόν 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, έτσι δεν είναι, α, εγκρίνεται, εγκρίνεται. Υπαριθμόν 3 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κύριε Γκουριάνου, παρακαλώ. Vote. Στο Πρόεδρε, μετά ψηφορία και σύμφωνα με τη θέση της ομάδας μου να προτείνω να υπερψηφίσουμε, να ψηφίσουμε υπέρ δηλαδή. Ευχαριστώ. Daraus schließe ich, dass die Einschätzung über die Άρα, είναι μάλλον απεσιόδειξη η πρόβλεψη σας για το είναι έκβαση της ψηφοφορίας, έτσι. Ναι, Πρόεδρε, και εμείς ε, περιμέναμε άλλη συμμετοχή στην ψηφοφορία. Κύριε Σαλαφράγκα. Όχι. Όχι. Άρα, ίσως θα έπρεπε να γίνει περισσότερη προσπάθεια με τις συμβαστικές τροπολογίες από ό,τι έγινε στην πράξη. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. Abstimmung ist ψηφοφορίας. 27 ψήφοι υπέρ, 26 ψήφοι κατά, εγκρίνεται η έκθεση. Ίσα ίσα. Κύριε Γκάλερς, δεν μου λέτε τέτοια τώρα. Και τώρα πάμε στην γνωμοδότηση Ρούσεκ, έτσι δεν είναι, πώς το προφέρουμε. Α, Ρότσεκ. Εδώ είναι. Στο ποδόσφαιρο έχει μείνει και αυτός. Κύριε Τσάλερ, έχετε τίποτα εσείς να μας πείτε, όχι. Λοιπόν, υπέρ της παριθμών 1 τροπολογίας, κατά, αποχές εγκρίνεται, ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο. Άρχεται. Πέρας. τα δύο υπέρ. Μετράμε.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 Meine Κυρίες και κύριοι, θέλω να τη συνεδρίαση. Ο κύριος Τζεντιλίνη και ο κύριος Μιρέλ είναι εδώ. Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Συζητάμε τις εξελίξεις στη Σερβία μετά τις εκλογές. κοινοβουλευτικές, δημοτικές, προεδρικές με αναπάντεχα αποτελέσματα. Οι διεθνείς παρατηρητές, έρατε και εσείς, έχουν πει ότι ήταν ε, καθαρές εκλογές, ανώθευτες. Με επιφυλάξω όμως ως προς τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη διαφάνεια. Δηλαδή κάποιες βελτιώσεις χωρούν ακόμη στο πεδίο αυτό ο πρόεδρος Νίκολετς είχε συναντήσει τον Φιούλε, τον κύριο Φαν την ε, κυρία Άστον πριν από τις εκλογές. Διεπίστωσε ότι η Σερβία είναι αποφασισμένη να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα τιμήσει κάθε συμφωνία που έχει να κάνει με το διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας και την υλοποίηση των ε, μεταρρυθμίσεων. Ε, επίσης, επισημάνθηκε ότι το Σύμφωνο σταθεροποίηση και Ανάπτυξη έχει κυρωθεί από όλες τις χώρες μέλη, πλην μίας. και θέλω να μάθω ποια είναι αυτή που δεν το έχει κυρώσει, για να μπορέσει να προχωρήσει σε ένα πολύ σημαντικό βήμα βέβαια της ε, ένταξης της ε, Σερβίας, ε, η οποία έχει αναπτύξει και καλές γειτονικέ σχέσεις με τους γειτονές της και θα πρέπει να τη στηρίξουμε στην προσπάθεια αυτή. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσεντιλίνη για πέντε λεπτά, μετά στον κύριο Μιρέλα, ο οποίος έχει πολλά να πει αλλά η φωνή του δεν τον βοηθάει. Έχει τεχνικές δηλαδή δυσκολίες ως προς το να σας μιλήσει. Γιατί έχει χάσει τη φωνή του. Κύριε Τζεντιλίνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά είμαι εδώ. Δύο λόγια θέλω να πω. Γιατί περιγράψετε πολύ σωστά το γενικό πλαίσιο η ενωσιακή μας πολιτική είναι πολύ σαφής για τη Σερβία και για την υπόλοιπη περιοχή. Έχουμε τα ουσιαστικά συμπεράσματα του Συμβουλίου των τελευταίων μηνών, τον, το Δεκέμβριο και το Φεβρουάριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, συζήτησε διαμακρών την διεύρυνση και πήρε αποφάσεις όχι μόνο για τη Σερβία αλλά για ό,τι την περιοχή για όλη την περιοχή. Και με αυτόν τον τρόπο δώσαμε ένα σαφέστατο μήνυμα ότι έχουμε σκοπό να προχωρήσουμε με την ατζέντα της διεύρυνσης. Υπάρχει η διεύρυνση στις συζητήσεις μας. Ο Πιέρ θα το αναπτύξει περισσότερο το θέμα αυτό. Ε, πρόκειται για την ατζέντα της Θεσσαλονίκη και έχει όλα τα στοιχεία εκτός από τα χρονοδιαγράμματα. Γιατί φυσικά αυτό εξαρτάται από την κάθε περίπτωση, πόσο γρήγορα προχωράει κάθε χώρα. Αλλά το βασικό είναι ότι θέλουμε ένα έντονο και θετικό μήνυμα στη Σερβία και στην περιοχή. Η περιφερειακή συνεργασία συζητήθηκε ως ένα πολύ σημαντικό σημείο. Σχέσεις δηλαδή με τις γειτονικέ χώρες είναι σημείο κλειδί και όταν δόθηκε, επάρθηκε η απόφαση να δώσουμε στη Σερβία την, το καθεστώς υποψήφιας χώρας, αυτό ελήφθη υπόψη. Τώρα θα έρθουμε στι εκλογέ, γιατί συζητάτε εδώ τι εκλογέ. Ο πρόεδρο υπενθύμησε τι συνέβη και ποια είναι η αποτίμηση των διεθνών παρατηρητών. Οι συζητήσει, όπω θα ξέρετε, για, την, για το σχηματισμό τη κυβέρνηση δεν έχουν ολοκληρωθεί και είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τι θα προκύψει από αυτέ τι συζητήσει. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Όσο, το συντομότερο, όσο συντομότερα σχηματιστεί η κυβέρνηση, τόσο καλύτερα. Ε, και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Ρωσίας. Όσο πιο γρήγορα έχουμε κυβέρνηση για να συζητήσουμε μαζί της, τόσο το καλύτερο. Αλλά αν είναι, υπάρχει κάτι που είναι γεγονός και μπορούμε να πούμε για την εκστρατεία και για τις ίδιες τις εκλογές, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ψηλά στη σερβική ατζέντα. Όλα τα πολιτικά κόμματα, τα βασικά πολιτικά κόμματα τα συζητάνε. Δεν είναι αμφιλεγόμενο θέμα, δεν αμφισβητήθηκε κάτι διάρκεια της προεκλογικής και και τα δύο βασικά, οι δύο βασικές παρατάξεις έχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προτεραιότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σημαντική η ατζέντα τους και εμπεριέχει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα χρειαστεί η Σερβία. Εμείς δεν ε, εμπλεκόμαστε σε αυτή την ε, πορεία. Όπως είπε και ο κύριος Μπλοκ, ο Μπροκ, ο Νίκολιτς είχε έρθει εδώ την περασμένη εβδομάδα και ήταν η πρώτη ευκαιρία για να συζητήσουμε α, τις σχέσεις με τη Σερβία, δηλαδή συμμετείχε και η Λέιδη Άστον, ε, μέσα σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα δηλαδή χώρα η συζήτηση και ήταν η πρώτη από πολλές συναντήσεις που θα λάβουν χώρα. Το μήνυμα ήταν ότι θέλουμε η Σερβία να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία και εμείς είμαστε στο πλευρό της Σερβίας. Φυσικά υπάρχουν διάφορα που πρέπει να γίνουν για το διάλογο. Ο Νίκολιτς είπε ότι θέλει όλες οι συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί να εφαρμοστούν. Και αυτό ήταν θετικό από πλευράς του. Και μόλις σχηματίστηκε η κυβέρνηση, όταν θα έχουμε την ευκαιρία, θα προχωρήσουμε ακριβώς αυτό. Μετά από αυτή τη συζήτηση που συζήτησε και τα θέματα συμφιλίωσης και περιφερειακής συνεργασίας μάθαμε ότι θέλει να συμμετάσχει η Σερβία σε αυτή την προσπάθεια, προσπάθεια να χυθεί φως στο παρελθόν και μετά από αυτή τη συζήτηση ο Ρόμπερτ Κούπερ θα πάει και στην Πριστίνα και στο Βελιγράδι αύριο γιατί θέλουμε να συζητήσουμε εν πάση λεπτομερία τη συμφωνία, σε τι φάση εφαρμογή βρίσκεται ποιος πρέπει να κάνει τι. Και νομίζω ότι αυτά αρκούν από την πλευρά μου. Ευχαριστούμε. Κύριε Μιρέλη, εσείς έχετε το λόγο. Ο πρόεδρος είπε ότι χάνω τη φωνή μου και θα δυσκολευθώ να μιλήσω, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Πριν έρθει ο κύριος Νίκολιτς ε, στις Βρυξέλλες στις 14, ο Επίτροπος Φίλε είχε προσκληθεί να παραστεί την, στην τελετή ανάληψη των καθηκών, δηλαδή ανάληψη των καθηκόντων του, ως πρόεδρος ε, της Σερβίας, εκλεγμένος πρόεδρος της Σερβίας. Και ή θα σχηματίσει η κυβέρνηση, θα είναι τμήμα της κυβέρνησης ο Νικόλιτς. Ε, έστειλε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα λοιπόν αυτό. Για τις σχέσεις με το Κοσφοπέδιο, να μην ε, πω αυτά που είπε ο Φερνάντο. Τα άλλα που είπαν ήταν για την περιφερειακή συνεργασία και τη συμφιλίωση στην περιοχή. Και κυρίως μετά από τις δηλώσεις που έκανε ο Νίκολιτς. Στις 15 Μαΐου είχαμε τη συνοκορυφής της SECP e στο Βελιγράδι όπου ο Νικολίτς επανέλαβε αυτά που είχε ήδη πει στις Βρυξέλλες. Ότι δηλαδή ήταν απόλυτα δεσμευμένο στην περιφερειακή συνεργασία και στην διαδικασία συμφιλίωσης. Ο Επίτροπος Φίλε έστειλε μια σειρά από σαφή μηνύματα που υπήρχαν και στην έκθεση πρόοδου του Οκτωβρίου ούτως ή άλλως και κάποια από αυτά αφορούν την σημαντική δικαστική μεταρρύθμιση, ότι θα πρέπει αυτή δηλαδή να συνεχιστεί και να εξασφαλίσει η Σερβία ότι οι δικαστές και οι... τι θα γίνει με τους δικαστές και τους εισαγγελείς. Τώρα, για την ελευθερία των ΜΜΕ, οι εκλογές έδειξαν ότι αυτή η ελευθερία μπορεί να βελτιωθεί πολιτική κατά της διαφθοράς. Πρέπει να γίνουν πολλά από αυτού στη Σερβία. Και το τελευταίο και σημαντικό μήνυμα είναι ότι χρειάζονται επιγόντως οικονομικές και διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή. Πέφτει η ισχύση του νομίσματος τις τελευταίες εβδομάδες. Γι' αυτό η χώρα χρειάζεται πολύ γρήγορα κάποιες σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Αυτά είναι τα μηνύματα που πέρασε ο Επίτροπος Φίλε και έδειξε τη διάθεσή μας να βοηθήσουμε σε όλα αυτά τα θέματα ανάλογα με τις ανάγκες της Σερβίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Κούγκαν που είναι πρόεδρος αντιπροσωπείας. Ο ένας δεν έχει φωνή και ο άλλος δεν έχει μικρόφωνο. Ναι, μια-δυο παρατηρήσεις, Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τους δύο μιλητές. Δεδομένης της σημαντικής θέσης της Σερβίας στην περιοχή, και της ε, διάθεσής μας να, να συνεχίσουμε με την ε, διεύρυνση. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε την ε, συνεργασία με τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο της Σερβίας, τον κύριο Νίκολιτς, και με την κυβέρνηση που θα σχηματιστεί μετά από αυτές τις ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. Πρέπει να κρίνουμε τον νέο πρόεδρο και τη νέα κυβέρνηση με βάση τα όσα θα πούνε, δεν θα πρέπει να το θεωρούμε κακό εκ των προτέρων, τον κύριο Νικολίτσο, όπως γίνεται σε ορισμένους κύκλους. Είναι δεσμευμένος να προχωρήσει με την περιφερειακή συνεργασία με σκοπό και την πλήρη ένταξη της Σερβίας στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει ο διάλογος ξανά Βελιγραδίου-Πριστίνας. Πρέπει να δούμε εμείς τι θέλουμε από αυτό το διάλογο και τι θέση θα κρατήσουμε στο μέλλον, γιατί ο πρόεδρος Νίκολιτς είπε ότι εκείνος θα πρέπει να είναι επικεφαλής στη διαπραγμάτευση από σερβικής πλευράς. Δεν μπορώ να φανταστώ τι μορφή θα πάρει αυτός ο διάλογος στην πράξη. Επίσης θα πρέπει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να, μιλάνε ομόφωνα. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Νικολίτς, ο, Ράμπουι, ο Φαρόμπουι, η Άστον και ο Μπαρόζο δεν είπαν πράγματα αντίθετα ένας προς τον άλλο. Φυσικά, οι εξελίξεις στο κοσφοπέδιο είναι πολύ σημαντικές. Δεν υπάρχει αναγνώριση της του κοσμοπέδιου της τη Σερβία. Το βασικό είναι να, να εξομαλυνθούν οι σχέσεις με το κοσμοπέδιο Ε, εμείς μιλούσαμε ε, μετά το 1968, όταν ε, έγινε η εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης, ε, μιλούσαμε για ε, εξομάλυση. Το θέμα είναι τι εννοούμε με αυτόν τον όρο εξομάλυση. Δηλαδή, σχέσεις που δεν θα υποσκάψουν τη σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων. Καλό θα ήταν βέβαια να ξέρουμε και το συγκεκριμένο περιεχόμενο της της εξομάλυνσης αυτής. Παρά να ακούμε, ας πούμε, μεγάλα λόγια, έτσι, θεωρητικά από καθέδρας για τον όρο αυτό. Αυτά. Ευχαριστώ. Κύριο Σόφλιν. Και από εδώ και πέρα θα ήθελα οι παρεμβάσεις να παραμείνουν στα δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι Συμφωνώ με αυτούς που παραδέχονται το γεγονό ότι ο Νίκολης εκλέχτηκε δημοκρατικά. Εγώ τον συνάντησα για μία ώρα τον Νοέμβρη. Η εντύπωσή μου είναι και δικιά μου και των άλλων στο Βελιγράδι ότι η δεσμευσή του Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ειλικρινής. Βεβαίω ενώπισα και το κόμμα του για αυτό το λόγο η υποδοχή λοιπόν της επιτυχίας του στα διεθνή ΜΜΕ νομίζω ήταν εσφαλμένη κατά την άποψή μου και θα έλεγα ότι όσον αφορά τις τελευταίες χειρονομίες και δηλώσεις του νομίζω υπάρχουν και άλλες πιθανές αναγνώσεις σε σχέση δηλαδή με την ανάγκη να καθησυχάσει τους ψηφοφόρους ο Νίκολιτς και η σερβική κοινωνία δεν σκέφτονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Γιατί ένα σημαντικό τμήμα τη σερβική κοινωνία ανησυχεί με την ευρωπαϊκή προοπτική και θα πρέπει να γίνουν και κάποιε χειραγωγήσει τέλο πάντων. Θα έλεγα λοιπόν ότι το κυριότερο πρόβλημα είναι η οικονομία που βρίσκεται σε κακή κατάσταση με υψηλά επίπεδα ανεργία, κυρίω μεταξύ των νέων, γύρω στο 50%, εξαρτάται πώ το υπολογίζει κανεί. Όσον αφορά τώρα την γενικότερη πολιτική, θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να φανταστούμε ότι κάποιος είναι λιγότερο εθνικιστής από τον Νίκολιτς. Ντάτσις, Βούτσις και άλλοι, όλοι είναι εθνικιστές, εξίσου με τον Νίκολιτς. Τη στιγμή που εξελίχθηκαν πολιτικά την εποχή του Μιλόσεβιτς, να μην το ξεχνάμε αυτό. Θα έλεγα λοιπόν ότι παραμένει αυτή πληγή και ο βομβαρδισμό τη Σερβίας που τραυμάσε τη σερβική κοινωνία. Δεν θα πρέπει να έχουμε μεγάλε προσδοκίε, και στο κάτω-κάτω θεωρώ ότι πολλά θα πρέπει να γίνουν ακόμα. Ακούσαμε τα διάφορα θέματα στη Μέση Διάταξη, ΜΜΕ, διαφθορά κλπ. Και κάτι άλλο σημαντικό. Θα πρέπει να υπάρχει όσο ευρύτερη γίνεται πρόσβαση στο ίντερνετ, ώστε να διασφαλίσουμε την ε, πολυφωνία απόψεων. Και επίση δεν θα απέκλεια το γεγονό ότι το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών να οδηγήσει σε μεγάλη κυβερνητική συμμαχία, αλλά τέλο πάντων θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Κόπα για δύο λεπτά. Uh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ για τι παρουσιάσει σα. Ο σωρικό λαό έκανε μια δημοκρατική επιλογή. Θα πρέπει να την αναλύσουμε σωστά και να τη σεβαστούμε. Κατά δική μου άποψη και τη ομάδα μου ο σερβικός λαός, η Σερβία γενικότερα δεν επέλεξε να εγκαταλείψει την ευρωπαϊκή προοπτική. Ο κ. Νικολής εκλέχθηκε με στενή, με μικρή πλειοψηφία και συμφωνώ θα πρέπει να δαιμονοποιήσουμε τον πρόεδρο Νίκολιτς. Έκανε αυτές τις ανησυχητικές δηλώσεις και πιο ανησυχητική από όλες αφορούσε τη γενοκτονία στη Σεβρενίτσα, κάτι το οποίο κατά την άποψή μας είναι μια υποχώρηση. Και χαιρόμαστε που ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς εξέφρασε την αγανάκτηση του σώματος την περασμένη εβδομάδα. Επίσης, θεωρούμε ότι η νέα Σεροκή Προεδρία θα πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά των προκατόχων της για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας, της σταθερότητας και της ειρήνης στα Βαλκάνια. Ξέρουμε ότι ο σχηματισμός κυβέρνηση είναι δύσκολο έργο από τη στιγμή που περιλαμβάνει πολλά κόμματα το Σερβικό Κοινοβούλιο. Χρειάζεται όμως συμβασμός περισσότερο από ποτέ και όλοι θα πρέπει να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα στο Βελιγράδι ότι θέλουμε μια λειτουργική κυβέρνηση να σχηματιστεί το ταχύτερο δυνατό κυβέρνηση που θα συνεχίσει τις ε, μεταρρυθμίσεις προς την ευρωπαϊκή ένταξη. Τέλος για τον Κωσυφοπαίδιο συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κούκαν ότι θα πρέπει ο διάλογος να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατό και η θέση μας για την εξουμάλυση των σχέσεων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα δεν συμμερίζομαι την απόψη του σε σχέση με την εξομάλυση ότι δηλαδή αποτελεί μια πολύ προχωρημένη στάση. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να έχουμε τέτοια προσέγγιση. Νομίζω θα είναι πολύ πιο εύκολο για την ε, Σερβία και για άλλες χώρες να γίνει κάτι τέτοιο οι η υπό την αιγύρα τη ευρωπαικη ενωση θα πρέπει να εφαρμοστούν, θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος και νομίζω ότι αυτή είναι μια διαδικασία που όλοι θα πρέπει να υποστηρίξουμε και όλοι γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια αυτη τη διαδικασια η Σερβία θα μπορούσε να προστατεύσει τα δικαιώματα των Σέρβων που διαμένουν στο Κόσοβο και βεβαιω θα μπορούσε να βοηθήσει μια τέτοια στάση την επίτευξη συμφωνια όπως και εμείς βεβαίως θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε ενεργά και να προστατεύσουμε τους, ε, τη συμφωνία και την ειρήνη εμείς. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Κονέλησον παρακαλώ. Θα είμαι σύντομη γιατί η κυρία Κοπά ήδη είπε πολλά από αυτά που θέλω να πω. Να ρωτήσω κυρίως κάτι σε σχέση με τα ατυχή σχόλια του κυρίου Νίκολιτς σχετικά με, την, ε, την γενοκτονία στη Σεβρενίτσα. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό ζήτημα. Άκουσα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι εντάξει αυτά είναι δηλώσεις αλλά νομίζω δεν θα πρέπει να απαβαίνουν αυτές τις δηλώσεις εις βάρος των ε, σχέσεων γειτονικών χωρών. Θα ήθελα λοιπόν να, ε, να μου πείτε τι θα κάνουμε με αυτό το ζήτημα και πώς θα το αντιμετωπίσουμε μελλοντικά. Ευχαριστώ κύριε Νίτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ένα αποσία του συναδέλφου Κακατσίν που είναι εισηγητής για την ε, Σερβία. Θα ήθελα να παρουσιάσω σύντομα την θέση της ομάδας μου. Ξέρετε ότι η ομάδα μου από την αρχή είχε μια κριτική υποστήριξη της, προς τη Σερβία για την προσχώρηση της δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγκαιρα χωρίς να είμαστε ενδοτικοί, τόσο πάμε κάποια αυστηρότητα σε σχέση με τα κριτήρια που θα πρέπει να πετύχει. Νομίζω ότι η εκλογή Σερβία ήταν αρκετά σωστές και διαφανείς, οπότε δεν ξέρω όμω με το γενικό αποτέλεσμα κατά πόσο θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Και δεν ξέρω τι γίνεται με την προσωπικότητα του εκλεγμένου Προέδρου. Πάντω, όπω και να έχουν τα πράγματα, θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί του. Και βεβαίω ε, λυπάμαι για τι δηλώσει του Προέδρου για τη Σεμπρενίτσα ότι εκεί δεν είχαμε γενιοκτονία. Νομίζω ότι ήταν ασφαλμένη η δήλωση και η τοποθέτηση αυτή. Νομίζω θα πρέπει να πούμε ότι έχει τεράστια σημασία ότι θα πρέπει να εξομαλυθούν οι σχέσεις μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Βεβαίως για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, αλλά επειδή επίσης φαίνεται ότι το βόρειο Κωσυφοπέδιο φαίνεται να αποτελεί μια όαση εγκληματικών δραστηριοτήτων στην ε, περιοχή και αυτό δεν είναι καλό. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση ώστε να υπάρξουν περισσότερες αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος. Βάγγελ. Ευχαριστώ. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα των εκλογών στη Σερβία ήταν ότι το συντηρητικό τμήμα της σερβικής κοινωνίας και πολιτικών ε, είχαν ευκαιρία να συμμετάσχουν και να, αναλάβουν και την ευθύνη για το ευρωπαϊκό μέλλον της Σερβίας. Θεωρώ ότι η εκλογή του Νίκολιτς ότι δεν είναι και τόσο άσχημη, άσχημα νέα. Δεν πρέπει να βάζουμε όλα τα αυγά σε ένα καλάθι και να ελπίζουμε ότι ο Τάντιτς και εκείνοι που ήταν ηγέτες της χώρας στο παρελθόν ε, είναι η μόνη μας χώρα, η μόνη, είναι η μόνη ελπίδα της Σερβίας. Συγγνώμη. Φυσικά οι αρχικές δηλώσεις του Νίκολιτς ήταν ατυχείς και απεικονίζουν το γεγονός ότι είχε μια τοπική εμβέλεια, δεν είχε διεθνή εμπειρία, ούτε είχε επαφές ποτέ μέχρι τώρα με πολιτικούς στην Ευρώπη. Από εδώ και στο εξή είμαι σίγουρος ότι θα λάβει υποστήριξη από τους Ευρωπαίους συντηρητικούς, το χρειάζεται. Ούτως ή άλλως οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί έχουν υποστήριξη και χειρότερος από αυτόν. Φυσικά υπάρχουν κάποια λεπτά θέματα. Μιλάω για τις θέσεις του Νίκολιτς. Το ένα είναι το κοσφοπέδιο και το άλλο είναι η Βοσνία και, η Βοσνία Η δήλωση της Στρεμπενίτσα παραπέμπει στον Ντόντικ. Αυτό δεν, είναι, δεν ήταν σωστό, ούτε υγιές. Φυσικά τα οικονομικά προβλήματα της Σερβίας είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσει η Σερβία να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αλλά έχουμε ένα καλό παράδειγμα στη Βοηγοντίνα. Πρέπει να εκτιμήσουμε, να συνεκτιμήσουμε τις θετικές εξελίξεις στην Βοηγοντίνα. Όταν ξεκινάει κανείς με τα, χειρότερα, ε, οτιδήποτε συμβεί από εκεί πέρα φαίνεται πρόοδος, εξέλιξη, θετικά νέα κτλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κύριος ε, Κράις Ντόρφλερ. Συμφωνώ κατά 90% με τα όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Υπάρχει ένα πράγμα που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή μας Ένωση δεν είναι στην καλύτερη δυνατή της φάση. Αν κοιτάξτε τα διάφορα κράτη-μέλη, ακόμα και το δικό μου, τη Γερμανία, έχουμε δημόσιες συζητήσεις που με φοβίζουν. Δεν χρειάζεται να ακούσω τον κύριο Νίκολιτς για να φοβηθώ δηλαδή. Από πολιτικούς με φοβίζουν και άλλοι πολιτικοί από άλλες χώρες. Κοιτάξτε τι γίνεται ε, στην ε, Ουγγαρία, το Φίντε στην Ουγγαρία, κοιτάξτε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Το σημαντικό για τη Σερβία δεν είναι η ευρωπαϊκή της προοπτική. Το βασικό είναι οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται για τους δικούς της τους πολίτες ούτως ή άλλως η ένταξη δεν θα πρέπει να είναι το κίνητρο για τις μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσει για το συμφέρον του λαού. Πρέπει να υποστηρίξουμε τη Σερβία σε αυτόν τον αγώνα για μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσει είναι πάντα πιο επιτυχεί αν θέλεις να μεταρρυθμίσεις, να αλλάξεις, να μετασχηματίσεις τον εαυτό σου. Ο σκοπό δεν είναι το, το βασικό εδώ. Είναι η πορεία, είναι τα μέσα, τα διάφορα βήματα που θα περάσουμε. Αυτά που έλεγε ο Μπερλουσκόν ακόμα μου φαίνονται ας πούμε ανατριχιαστικά. Και αυτά που έλεγε ο κύριος Σαμαράς στην Ελλάδα, όταν κατέστρεφε την Ελλάδα, την ε, κυβέρνηση, την προηγούμενη. Ο κύριος Νίκολς δεν είναι ο μόνος ο οποίος λέει φρικόδη και ανατριχιαστικά πράγματα. Ας σκεφτούμε όλοι και ας κάνουμε ας πούμε, έτσι, μια αυτοκριτική για τους δικούς μας πολιτικούς. Φυσικά, η προοπτική για την ένταξη είναι πολύ σημαντικό πράγμα για τη Σερβία, αλλά θα χρειαστεί χρόνο. Εντάξει, οι εξέλιξει όντω κινούνται με ταχύ ρυθμού, αλλά αν κοιτάξετε πώ εξελίχθηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί αλλάξαμε άρδιν. Αλλά αυτέ οι αλλαγέ έγιναν μέσα σε μεγάλη χρονική περίοδο. Χρειάζεται δουλειά και υπομονή. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τάνοκ. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι φίλο τη Σερβίας και της ε, ευρωπαϊκής και ατλαντικής προοπτικής της. Δεν φαντάζομαι ότι στο εγγύς μέλλον θα ανταχθεί στο ΝΑΤΟ για προφανείς λόγους. Αλλά σύμφωνα με τον Κούκαν ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε τον νέο πρόεδρο τον Νίκολιτς. Η άρνηση της γενοκτονίας της Σεμπενίτς από μέρους του φυσικά ηθικά είναι ε, απαράδεκτη. Ε, σημαίνει ότι είναι αδαής ο άνθρωπος και δεν βοηθάει την ειρήνη και την συμφιλίωση στην περιοχή κύριος Σόφλιν ανέφερε την ε, οικονομία. Αλλά το 50% των νέων που είναι άνεργοι στη Σερβία ε, δεν είναι μεγαλύτερο αυτό το ποσοστό από ότι στην Ισπανία, ας πούμε, ή αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, με ενδιαφέρουν οι σχέσεις με το Μαυροβούνιο, γιατί είμαι ο εισηγητής του Κοινοβουλίου για το Μαυροβούνιο. Νομίζω ότι οι σχέσεις πάνε καλά. Αλλά φαντάζομαι ότι οι... κάποιοι από τους εθνικιστές δεν αρέσκονται σε αυτό το διαχωρισμό στο βάθος της καρδιάς τους. Ελπίζω να συνεχίσει ο Νίκολης τις ε, καλές σχέσεις με το Μαυροφούνιο για το κοσφοπέδιο. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να βάλουμε όλες τις εναλλακτικέ λύσεις επιτάπητος εμείς οι δυτικοί. Ε, ε στην πραγματικότητα φτιάξαμε μια κατάσταση που είναι ανεπίλητη εις βάρος του Ευρωπαίου φορολογούμενου και εμείς και οι Αμερικάνοι μαζί. Έχουμε το οργανωμένο έγκλημα, όχι μόνο στο Κοσμοπέδιο βέβαια, αλλά σε όλη την περιοχή δυστυχώς. Επίσης, ε, βόρεια του ποταμού ε, Μπαρ ε, είναι μια χώρα που δεν σε κανένα no man's land. ελπίζω να επιληθεί το πρόβλημα αυτό σύν το χρόνο. Ο κύριος Λανσμπέργκης. Η ερώτησή μου είναι η εξής είναι γεωπολιτική για την ε, Σερβία. Υπάρχουν ενδείξεις ή όχι ότι η Σερβία ε, διολυσθένει προς μια κατάσταση προτεκτοράτου της, Σερβία, της ε, Ρωσίας. Νομίζω ότι τα κατάφερε η Ρωσία. Ε, τα κατάφερε και σε αυτή την περιοχή. Τα ίδια έγιναν και στην ε, Λιθουανία. Ε, προωθήθηκαν οι υποψήφοι της Ρωσίας. Η Ρωσία είναι ακόμα πολύ σημαντική και έχει επιρροή. Αυτή η συμμαχία Ρωσίας-Σερβίας ήταν ακόμα μια φορά καταφανής. Όπως ε, την περίοδο των ατυχών πολέμων του Μιλόσεβιτς. Εγώ αυτό πιστεύω. Εσείς τι στοιχεία έχετε. Ο κύριος Πίκουλα. Thank you. As the Ευχαριστώ. Ως παρατηρητής στις σερβικές εκλογές πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι ήταν σαραστημένοι από το προηγούμενο πρόεδρο γι' αυτό δεν τον ψήφισαν. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι δεν θέλουν να έχουν κακές σχέσεις με τους ε, γειτονές τους είχαμε περισσότερο κοινωνικά διλήμματα και ζητήματα που υπερίσχυσαν. Θα πρέπει νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει τις πόρτες ανοιχτές, τις πόρτες για τη Σερβία και για άλλες χώρες των ε, Δυτικών Βαλκανίων, αλλά θα πρέπει να αφήσουν φαντάσματα να πέρασουν από αυτές τις πόρτες. Γενικά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει έναν μεσολαβητή επιτυχημένο στα Βαλκάνια, όπως ακριβώς έκανε στην ε, Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Η Κροατία έχει και αυτή μεγάλο ενδιαφέρον και συμφέρον να δει την Σερβία, το Βελγάρα να προοδεύει προς την Ευρώπη. Αλλά βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από σημαντικές διαφορετικές αλλαγές που θα αποτελέσουν και άλλα μέτρα που θα αποτελέσουν ένα σημαντικό δίκτυ σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Γκόμες. Οι συνάδελφοι Κόπα και Κράση Τέφλερ ήδη έκαναν την ίδια ανάγνωση που έχω και εγώ. Να πω μόνο ότι Συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Πίκολα μέχρι τώρα. Οι ψηφοφόροι στη Σερβία επηρεάστηκαν από τις επιπτώσεις της δικής μας κρίσης στη Σερβία. Περί αυτού πρόκειται. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν πώς θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να τους δώσει περισσότερα επιχειρήματα και κίνητρα στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο για να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο μπορούσε να ήταν περισσότεροι αποτελεσματικοί στην πρόσληψη αυτών των κινήτρων στην κοινωνία των πολιτών. Ίσως η ηγεσία να είναι λίγο αφήσιμη καμιά φορά, αλλά πώς θα μπορούσαμε να εμπλέξουμε την κοινωνία των πολιτών στη Σερβία και, ώστε να κατανοήσει ότι το, μέλος, το μέλλον τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε επίσης διαρωτώ με την σερβική οικονομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Τζεντιλίνη και μετά κύριο Μίρεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να σχολιάσω δύο-τρία πράγματα που σχετίζονται περισσότερα με τη δικιά μου τη δραστηριότητα. Καταρχάς για το στόχο. Σε τι στοχεύουμε. Η σαφήνεια είναι πρακτική και φιλοσοφική, ενιολογική. Λοιπόν, μιλάμε για την εταιρική σχέση. Δεν μιλάμε για την αναγνώριση κλπ. κλπ. Η σχέση, η εταιρική σχέση. Και αν κοιτάξουμε τη δουλειά των περασμένων μηνών, ο διάλογος, οι συμφωνίες που κάποιες εφαρμόστηκαν, άλλες όχι, αλλά τέλο πάντων δεν είμαστε όλοι με την πρόοδο, αλλά αν κοιτάξουμε το πράγμα σφαιρικά, θα δούμε ότι θέλουμε να προοδεύσουμε στη συνεργασία, να βοηθήσουμε το λαό και να αφαιρέσουμε τα εμπόδια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια λειτουργική εταιρική σχέση και έτσι θα πρέπει να το προσεγγίζουμε το θέμα. Περιφερειακή συνεργασία. Βεβαίω και αυτή είναι πολύ σημαντική, για τη δήλωση επί ευκαιρία για την Σεμπρενίτσα. Νομίζω θα πρέπει να κάνουμε και γραπτή δήλωση και ήμασταν σαφείς και ξεκάθαροι από την αρχή. Είπαμε ότι δεν είμαστε εδώ για να ξαναγράψουμε ιστορία κλπ. κλπ γιατί βεβαίως τα γεγονότα σημαντικά, εξίσου και δηλώσεις και γι' αυτό ακριβώς ήταν σωστό να αντιδράσουμε αμέσως με σαφή τρόπο. Για τα γεωπολιτικά ζητήματα, είπα και προηγουμένως, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της Σερβίας και όσο πιο ξεκάθαρο είναι αυτό, τόσο πιο εύκολα θα είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία νομίζω από αυτού. Αυτά είχα να πω. Θα δώσω το λόγο στον Πιέρ. Ναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς για τις παρατηρήσεις της κυρίας ε, Κόπα και της Κονέλησεν για τη δήλωση σχετικά με την Σεμπρενίτσα. Όταν είχαμε συναντήσεις και στο Βελιγράδι και στις Βρυξέλλε με τον κύριο Νίκολιτς είπε ότι είχαν παρεμεινευτεί οι δηλώσεις του και λοιπά. Να πω όμως ότι από την αρχή και στο Βελιγράδι στην ε, τελετή ενάρξης και εδώ με Ρομπάι, Άστον, ...Μπαρός όπως είπε ο κύριος Κουγκάν όλα τα θεσμικά όργανα μιλούσαν με την ίδια γλώσσα δηλαδή συμφιλίωση περιφερειακή συνεργασία και προσέξτε τι λέτε. Αυτό ήταν το σημαντικό μήνυμα που έπρεπε να στείλουμε και που στείλαμε από την αρχή. Μετά λοιπόν αυτές τις σαφείς εξηγήσει, αν μπορώ να το πω έτσι, και να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Κούκαν ότι τους επόμενους μήνες θα κρίνουμε τι θα κάνουν. Και συμφωνώ με έναν άλλο ομιλητή όμως ότι ο κύριος Νίκολιτς ήδη έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο αν κοιτάξουμε το κόμμα του και την πρόσφατη πορεία του. Και απλά και μόνο το γεγονό ότι στην ε, τελετή έναρξη, μάλλον στην ανάληψη των καθεκόντων του και εδώ στις Βρυξέλλες μετά στη συνέχεια εξέφρασε την σαφή βούλησή του για την ανάπτυξη των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα να το λάβουμε, αλλά με πόσο μας ότι αυτό προέρχεται αμέσω μετά την εκλογή του για τη σχέση τώρα με το Μαυροβούνιο. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να θεωρούμε ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα και λόγω του γεγονότος ότι ο πρόεδρος του Μαυροβούνιου ήταν ε, από τους λίγους που παραβρέθηκαν στην, ανα... στην τελετή ανάπτυξη καθηκόντων κ. Νίκολης τον Ιούνιο. Για τα σχόλια τώρα, για την εκλογική εκστρατεία κλπ. Νομίζω ότι αυτοί που λένε Νομίζω κυρία Γκόμες το πει συγκεκριμένα ότι οι πολίτες δεν ψήφισαν βάσει εξωτερικής πολιτικής ή σχέσης με το κοσφοπέδιο, ψήφισαν ε, με κριτήριο άλλα στοιχεία, πιο καθημερινά όπως υψηλή ανεργία κλπ. κλπ. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ήταν χαμηλά προτεραιότητες τις εκλογικές το κοσφοπέδιο και εμείς είπαμε και ο κύριος Φίλε ανέφερε και επανειλημμένα υπόθηκε ότι υπάρχει ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στη Σερβία που θα αφορούν τον αντογανισμό επειδή έχουμε πολλά μονοπόλια που διατηρούν τις τιμές υψηλές, διαφορετικές αλλαγές, ιδιωτικοποιήσεις, μεταρρυθμίσεις που αφορούν τα ΜΜΕ κλπ. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να βοηθήσουμε αλλά βεβαίως αναμένουμε και την αντίστοιχη βούληση η ανάληψη αυτών των μεγάλων μεταρρυθμίσεων ώστε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Νομίζω πάντως οι γενικέ γραμμές δεν θα πρέπει να υπάρχει αφιβολία και εσείς το γνωρίζετε καλά ως σώμα ότι είναι προς το συμφέρον όλης της περιοχή και της Ευρώπης γενικότερα να προχωρήσει και να προσχωρήσει η Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Τζαντιλίνη, κύριε Μιρέλ, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφου. Στις 10.30 θα συζητήσουμε το επόμενο σημείο μας, ε, όταν θα έρθουν όλοι οι προσκεκλημένοι μας. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι τις 10.30. Συνεχίζουμε με το επόμενο σημείο στην μέση διάταξη. Δραστηριότητα του Εθνού Ποινικού Δικαστηρίου στη Λιβύη. Καλώ ορίζω την κυρία Σφαλ Κόρμαν και την κυρία Τζένιφερ Σέντ, σύμβουλο για τη Διεθνή συνεργασία. να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω την 9017 απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που μιλάει για το θέμα του εισαγγελάτου του Εθνούς Δικαστηρίου στη Λιβύη και να επενθυμίσω ότι η Λιβύη δεν έχει ακόμα αναγνωρίσει το ρόλο του και ζήτησε το Κοινοβούλιο να το κάνει αυτό στα πλαίσια της ε, συμφωνίας που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Λιβύη. Να επενθυμίσω επίσης ότι η πρόσφατη απόφαση Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Λιβύη εκφράζει σημαντικές ανησυχίες για παράνομες κρατήσεις, βασανισμούς, εκτελέσεις στη Λιβύη και καλεί να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της παραβίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λιβύη έχουμε και το θέμα του Σαΐφ και του Απτουλά Σαντούση που αποφάσισε η Λιβύη να τους ε, δικάσει και υπάρχει έτοιμα διεξαγωγής έρωνας και εκδίκαση των υποθέσεων αυτό από το διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Θεωρεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε αυτή την περίπτωση έχουμε σαφείς παραβιάσεις και παρακολουθεί στενά τις υποθέσεις αυτές και ζητείται η άμεση απελευθέρωση όπως αναφέρει και η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιουνίου. ώστε να έχουν ελευθερία οι κρατούμενοι και να έχουν ελευθερία επαφή με τις οικογένειές τους και να έχουν μια δίκαιη δίκη. Καλωσορίζω λοιπόν την κυρία Σπαρκόπαν, η οποία θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις εδώ στην Επιτροπή μας. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να έρθω εδώ σήμερα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας για την κατάσταση στη Λιβύη. Είναι μια καλή ευκαιρία αυτή για μας και επιτρέψτε μου να πω καταρχάς ότι είμαι ευγνώμων για την σημαντική υποστήριξη που είχαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γενικότερα της ε, υπηρεσίας του δικαστηρίου, αλλά και συγκεκριμένα του Σαγγελέως. Ήταν μια από τις πιο σημαντικές υποστήριξεις που είχαμε, ιδιαίτερα μετά από την έκθεση του Απρίλη που δημοσιεύσαμε. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη δουλειά μας. Εσείς μας υποστηρίξατε για την ε, σύνταξη ενός ε, κώδικα δεοντολογίας και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί ξέρετε ότι κράτη και οργανισμοί θα πρέπει να επιτρέπουν τις επαφές με τους κρατούμενους. Έχουμε το θέμα επίσης των ε, θαντικών ε, ποινών και το θέμα της ρήτρας με τις συμφωνίες σε με τρίτες χώρες και βεβαίως το θέμα της προστασίας αυτής της ε, ρήτρας της συμφωνίας με τρίτες χώρες είναι πολύ σημαντική για μας. Με χάρα επίσης είδαμε την αναφορά στην χρηματοδότηση για το δικαστήριο. Αυτό αποτελούσε μια ανησυχία ε, για μας, μας ανησυχούσε και το αναφέραμε στις συζητήσεις τον περασμένο Δεκέμβρη και μας ε, καθυσυχάζει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την σωστή χρηματοδότηση του δικαστηρίου, στο αυτό να εκτελέσει την εντολή του. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και πάλι για τη σημαντική ε, υποστήριξη προ εμά. Αν συμφωνείτε λοιπόν, θα παρουσιάσω σε λίγα λεπτά την κατάσταση στην Λιβύη και μετά συνάδελφο και εγώ θα απαντήσουμε ευχαριστώ σε ερωτήσει σα λεπτομερεί. Και όπω ανέφερε και ένα συνάδελφο, το Συμβούλιο Ασφαλείας συζήτησε την κατάσταση Λιβύη το 2011 με συνένεση και αυτή η συνένεση ήταν πολύ σημαντική για μας γιατί μας επέτρεψε να έχουμε μια αυξημένη συνεργασία. Είχαμε λοιπόν πολύ καλή συνεργασία και αυτό μας επέτρεψε να προχωρήσουμε γρήγορα. Μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε μια προκατακτική εξέταση και να ξεκινήσουμε δικασία εξέτασης πολύ σύντομα και να αναλάβουμε και την πρώτη υπόθεση. Αυτό ήδη το κάναμε από τον Μάιο. Κατά τριών ατόμων, Μουαμαρ, Σασαΐφ και τον επικεφαλής της ε, μυστικής ε, αστυνομίας των Σαούση. Είχαμε λοιπόν περιπτώσεις παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φόνος, δολοφονίες κλπ. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι εδώ δεν εξετάζουμε μόνο όλα τα εγκλήματα που διέπραξαν οι λιβικές αρχές κατά διάρκεια του καθεστώτος Καντάφη. Εμείς κοιτάξαμε λοιπόν μόνο αυτά που έγιναν από το Φλεβάρι του 2011. Επειδή λοιπόν είχαμε αυτή την συνεργασία μπορούσαμε να προχωρήσουμε γρήγορα και εξετάσαμε τα εγκλήματα που έγιναν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που σας ανέφερα. Μπορούσαμε λοιπόν πολύ γρήγορα να εξετάσουμε τις ε, κατηγορίες αυτές και είχαμε μια πρώτη απόφαση και έκδοση εντάλματος σύλληψης για αυτά τα τρία άτομα. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχουν παρκή λόγοι να πιστεύουμε ότι μετά από την Αραβική Άνοιξη του 2011 οι Λιβικές Αρχές ε, δημιούργησαν ένα σχέδιο καταστολής των αντιφρονούντων και χρησιμοποίησαν όλα τα μέσα για να καταστήλουν όλες τις διαδηλώσεις και τις εκδήλωσεις αντίθεσης και όπου δηλαδή συμμετείχαν οι αντιφρονούντες. Είχαμε λοιπόν συγκεκριμένα επιθέσεις. Θεωρούσαμε ότι αυτό αποτελούσε μάλλον επίθεση κατά του πληθυσμού, κατά των πολιτών της χώρας. Ο Ασίφ ε, συνελήφθη στο Σιντάν και οι νέε λιβικέ ε, αρχέ μα είπαν ευχαριστούμε πολύ Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο για την δράση σα, για την ε, υπογράμμιση και την έμφαση στο ρόλο τη ε, της δημοκρατίας στην περίπτωση αυτή, αλλά θα θέλαμε να το χειριστούμε μόνοι μας. Εμείς όμως έχουμε ένα συγκεκριμένο καταστατικό που μας υποχρεώνει να δράμε ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και βεβαίως εμείς ε, ως δικαστήριο και οι δικαστές θα πρέπει να δεσφαλίζουμε την εφαρμογή τη της μα όπου υπάρχουν ε, εθνικές διαδικασίε, αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται. Είπαμε λοιπόν ξεκάθαρα στι ελληνικέ αρχές ότι θα πρέπει να εφαρμόσουν τις διαδικασίε αυτές και έλαβαν υπόψη του σοβαρά αυτά που τους είπαμε, κοίταξαν και το καταστατικό και έχουμε ένα λεπτομερές έγγραφο ως αποτέλεσμα το οποίο εξηγεί στην ουσία ότι ο Γενικός Εισαγγελέας στην Λιβύη κάνει έρευνα για τον Σαΐφ για κάποια σοβαρά εγκλήματα που διαπράχτηκαν κατά διάρκεια της εξέγησης του 2011 από το Φλεβάρι μαζί με αυτά που έγιναν από το Φλεβάρι μέχρι το Μάη. Έχουμε λοιπόν τα ίδια εγκλήματα τα οποία εξετάσουμε και εμείς και είναι πολύ συγκεκριμένο το πλαίσιο στο οποίο δράμε. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με τα ίδια άτομα και τις ίδιες κατηγορίες. Είπαμε λοιπόν στις λιβικές αρχές ότι εξετάζουμε και ερευνάμε τις ίδιες υποθέσεις που ερευνάτε κι εσείς, οπότε όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται με συντονισμένο τρόπο και σύμφωνα με το καταστατικό. Είπαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεργαστούν λιβικές αρχές και θα πρέπει να τηρούν και να σέβονται τις διατάξεις ε, του καταστατικού, που όχι όπως το Σουτάν που λέει ότι δεν ε, συμφωνούμε με αυτό το καταστατικό, δεν τον τηρούμε, δεν το σεβόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να το τηρήσουν, να σεβαστούν το καταστατικό που αφορά τη δική μας δράση Αυτό λοιπόν δεν ισχύει εδώ. Χρησιμοποιούν οι ίδιε ελληνικέ αρχέ τι διατάξει αυτού του καταστατικού και στο τέλο θα πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι δικαστέ κατά πόσο θα πρέπει να γίνονται ουσιώδει και πραγματικέ δικαστικέ έρευνε. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε βεβαίω την ε, ε, σωστή διατροφή των κρατουμένων, την υγεία του. Θα πρέπει να έχουμε ε, και την εφαρμογή ψηλών προδιαγραφών όσον αφορά τι δικαστικέ έρευνε και όπως ζητήθηκε από τις συμμετέχοντες στην ε, ακροματική διαδικασία θα πρέπει να έχουμε και δυνατότητα απάντησης. Πρέπει τώρα λοιπόν οι δικαστές να αποφασίσουν, να εξετάσουν πολύ προσεκτικά την υπόθεση αυτή που είναι αρκετά που αποτελεί μάλλον μια πρόκληση. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, όταν αποδεχτήκαμε την υπόθεση αυτή, δεν εξετάσαμε το σύνολο του δικαστικού συστήματος της Λιβύης δηλαδή κατά πόσο είναι σε θέση το σύνολό του να ανταποκρίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά κοιτάξτε με συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως γνωρίζετε επίσης, ο Αλσανούση συνελήφθη στην Μαυρετανία. Η Μαυρετανία όμως δεν είναι χώρα μέλος. Μεταβιβάσαμε το αίτημα για την έκδοση του κατηγορούμενου και οι αρχέ λοιπόν τη Μαυρετανίας θα πρέπει να αποφασίσουν το πώ αντιμετωπίζουν αυτές τις, αυτά τα αιτήματα. Και η αλήθεια είναι ότι ο Αλτσανούση είναι ασθενή, οπότε δεν είχαμε κάποια εξέλιξη μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει και πάλι να αποφασίσουν οι αρχέ τη Μαυρετανίας τι θα κάνουν σε αυτή την υπόθεση. Επίση, ε, προχωράμε στην δεύτερη υπόθεσή μα. Δεύτερη υπόθεση, μαζί με αυτέ τι τρει αυτά τα τρία άτομα που σα ανέφερα, αφορά εγκλήματα κατά του φίλου συγκεκριμένα κατά γυναικών, σε συγκεκριμένες περιοχές της Λιβύης. Προσπαθούμε λοιπόν να συλλέξουμε στοιχεία τα οποία δεν επιφέρουν κινδύνους για τα θύματα μέσω γιατρών, μέσω στρατιωτών, μέσω, από, μέσω άλλων πηγών επίσης. Επίσης διερευνούμε και την ύπαρξη και άλλων υπόπτων του καθεστώτος ε, κατάφη που διαμένουν στο εξωτερικό Έχουμε λοιπόν διάφορες υποθέσεις αυτού του είδου που εξετάζουμε ταυτόχρονα. Γνωρίζετε επίσης έχουμε και μια εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ που έκανε μια έκθεση τον Μάρτι και που παρουσιάζει συνοπτικά τα εγκλήματα που έγιναν στη Λιβύη και που, και που έχουμε παραβίαση ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων, αλλά για την περίπτωση γενοκτονίας δεν ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα, γιατί το, η εντολή μας δεν είναι αρκετά περιορισμένη γι' αυτό. Έχουμε επίσης χιλιάδες άτομα τα οποία κρατούνται και υπάρχουν βεβαίως και κατηγορίες για κακομεταχείριση και βασανισμό αυτών των ε, κρατουμένων και εξετάζουμε και αυτές τις υποθέσεις. Επίσης καταγράψαμε και τα ευρήματα της Εξεταστικής Επιτροπής για την δράση του ΝΑΤΟ στην Λιβύη και εξετάσαμε και το κατά πόσο οι πολίτες αποτέλεσαν στόχο του ΝΑΤΟ στη Λιβύη, είχαμε πάρα πολλές αεροπορικές επιδρομές στη Λιβύη. Το σημειώσαμε λοιπόν αυτό. Εξετάσαμε πέντε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου προσπαθήσαμε να συλλέξουμε στοιχεία για να δούμε κατά πόσο είχαμε ένα θέμα Αναλογικότητα. δηλαδή κατά πόσο θα έπρεπε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να αποτραπούν οι απώλειες αμάχων μετά από αυτές τις επιδρομές. Η βάση μας είναι το 90 απόφαση. Δεν έχουμε λοιπόν την δυνατότητα να, να διερευνήσουμε την η ίδια τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ που αφορά άλλη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλεία, το ίδιο δηλαδή όπω και για την περίπτωση γενοκτονία όπου έχουμε περιορισμένη εντολή. Η κυβέρνηση τη Λιβύη κατανοεί τη σοβαρότητα αυτών των υποθέσεων και συντάξαμε ένα σχέδιο συνολικό για την αντιμετωπίση, για την αντιμετωπίση αυτών των υποθέσεων. Θα πρέπει βεβαίω να υπάρχει και απόδοση λογαριασμών, θα πρέπει να υπάρχει ανάληψη ευθύνη και θα πρέπει σε κάποιε περιπτώσει, για κάποιου κρατώμένου. θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να γίνουν συλλήψει ή κατά πόσο θα πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι άλλοι κρατούμενοι. Ζητήσαμε λοιπόν από τις εθνικές αρχές να αντιμετωπίσουν σοβαρά και αυτέ τι κατηγορίε για βασανισμούς και κακομεταχείριση των συλληφθέντων. Το κάνουμε αυτό βεβαίω σε όλε τι επαφέ που είχαμε με τι λιβικέ αρχέ και μα είπαν ότι έχουν στα σκαριά ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων. Μα είπαν επίση ότι θα ακολουθήσουν τι ίδιε πολιτικέ που ακολούθησαν για, τις, για τα πιο σοβαρά εγκλήματα, για τους κατηγορούμενους δηλαδή για τα σοβαρότερα εγκλήματα και για τις άλλες ε, περιπτώσεις θα προβλέψουν ένα είδος ε, μεταβατικού σχεδίου για την απόδοση της δικαιοσύνης μέσω μιας ε, επιτροπής εξεταστικής. Είναι σημαντικό λοιπόν να προσπαθήσουμε να τους ενθαρρύνουμε σε αυτή τη διαδικασία και έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή σε σχέση με την κατάσταση στη Λιβύη. Στη Λιβύη. Και πριν να κλείσω θα ήθελα να πω ότι σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη για κάποιους συναδέλφους που συλλήφθηκαν και είμαστε σε επαφή με τις λιβικές αρχές για την λύση οποιοδήποτε παρεξηγήσεων ώστε να απελευθούν συνάδελφοι το ταχύτερο δυνατό και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη μας όσο για τα θέματα αυτά. Η Τζένιφερ και εγώ είμαι εδώ για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία μας όσο να είμαστε εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, ευχαριστώ για την επισκόπηση. Θα ήθελα να αρχίσω με, με τις ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Η κυρία Γκόμες που είναι η συγγήτρια για τη Λιβύη ε, έχει το λόγο. Μόλις ήρθα από τη Λιβύη. Ε, υπάρχει εδώ και άνθρωπος που έχει επαφές με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Σε ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι συμπίπτουν αυτά που μα είπατε με τι πληροφορίε που έχω εγώ για τη Λιβύη, ότι οι λιβυκές αρχέ θέλουν να συνεργαστούν με το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο, ε, να σεβαστούν όλα τα στοιχεία που είπατε, θέλουν να δώσουν προτεραιότητα όχι μόνο στι πιο σοβαρέ ε, περιπτώσεις, στις πιο σοβαρές υποθέσεις, αλλά θέλουν να εγγύψουν και στο πρόβλημα των κρατουμένων. Το πρόβλημα είναι ότι το κράτος ε, στην Λιβύη είναι δυσλειτουργικό. Είναι η κληρονομιά του Καντάφη και φυσικά η δικαιοσύνη είναι ένας από τους θεσμού που δεν λειτουργεί καλά. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια και το αναγνωρίζουν, πιστεύουν και το αναγνωρίζουν, θα αποφευθούν από τη συνεργασία με το Διεθνικό Δικαστήριο και τη διεθνή κοινότητα. Εδώ ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιτείνει τη συνεργασία της με τις Λιβικές Αρχές. Φυσικά είμαστε σε δύσκολη συγκυρία τώρα. οι μεταβατικές αυτές αρχές υπάρχουν, θα ακολουθήσουν ε, εκλογές, φυσικά. Ξέρουν πολύ καλά ότι είναι, η εντολή που έχουν λάβει είναι περιορισμένη χρονικά, δεν θα μείνουν αιωνίως. Ε, και βεβαίως ε, παράλληλα με τη δυσλειτουργία της δικαιοσύνης υπάρχει και η δυσλειτουργία του, των υπηρεσιών ασφαλείας. Ε, οι μόνες υπηρεσίε που λειτουργούν καλά στη Λιβύη είναι οι πολιτοφυλακέ. Δεν λειτουργεί η αστυνομία, δεν λειτουργούν διάφοροι ιδιοκτικοί μηχανισμοί και βεβαίω η πολιτοφυλακή της ΖΙΝΤΑ. Ζιντάν, που ήταν υπεύθυνη για την τελευταία φάση της εξέγερσης και την εκδίωξη του Καντάφη από την Τρίπολη έχουν υποστήριξη και σε κάποια υπουργεία και πρόσφατα ελέγχαν το αεροδρόμιο της ε, Τρίπολης και μετέφεραν την ε, εξουσία στις ε, διεθνείς δυνάμεις, αλλά, η... ουσιαστικά τους ξαναπέταξαν πίσω τον μπαλάκι, γιατί μόνο αυτοί ήταν σε θέση να ελέγξουν το αεροδρόμιο. Αυτό δείχνει ακριβώς τις δυσκολίες που υπάρχουν στη Λιβύη. Ε, και φαντάζεστε και τις δυσκολίες που έχει και η ομάδα του ποινικού δικαστηρίου, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Σε όλες τις επαφές μου και με τα νεοσχηματιστέντα ε, πολιτικά κόμματα, πάντα έθεσα το θέμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και με τους ε, δημοσιογράφους επίσης. Οργανώθηκε μία σύνοδος έτσι, ένα σεμινάριο ας πούμε για, την, για τους δημοσιογράφους ε, και εκεί το ανέφερα, αλλά το ανέφερα με πολύ διπλωματικό τρόπο γιατί έτσι πρέπει να υποθούν αυτά τα πράγματα. Πρέπει να καταλάβετε τις ανησυχίες των Λίβιων. Έχουν κάθε σεβασμό σε αυτούς τους θεσμούς και πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Ξέρουν ότι υπάρχουν τεράστια ποσά χρημάτων παγωμένα ή κάπου κρυμμένα, εν πάση περιπτώσει, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διάφορες σε διάφορους παράκτιους ε, παραδείσους που ελέγχονται από ανθρώπους του Γκαντάφη και υπάρχει και απειλή και φόβος ότι άνθρωποι σαν τον ε, Σαϊφ Αλισλάμ θα εξισιοδοτήσουν άλλους ανθρώπους εκτός της Λιβύης για να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα, όχι για τους ίδιους, αλλά και για να... ούτε βέβαια θα τα δώσουν αυτά λεφτά στο λιβικό λαό, αλλά για να συνομωτήσουν εναντίον του λιβικού λαού Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν πάρα πολύ και τη στάση του απέναντι στο Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Γι' αυτό εγώ ήμουν πάρα πολύ διπλωμάτης, επειδή ακριβώ μιλούσα και δημόσια. Ότι υπάρχουν παρεξηγήσεις και από τι δύο πλευρές. Το είπα αυτό. Είπα ότι δεν υπάρχει αρκετή ευαισθησία στι πραγματικέ ανησυχίε του λιβικού λαού. Και στο ευαίσθητο θέμα των, της πολιτοφυλακής της Ζιντάν που κρατούσαν και τον Σαϊφ, κρατούν τον Σαϊφ και που έχουν πραγματική εξουσία μεταξύ όλων των φορέων εκεί στη Λιβύη είναι τους πιο ισχυρούς. Αυτό που είπα δημόσια το λέω και εδώ μίλησα για αυτές τις παρεξηγήσεις είπα στους Λίβιους ομολόγους μου ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα ε, στην εικόνα της ε, Λιβύης στο εξωτερικό και στα ΜΜΕ. Αυτό δεν το αξίζει η Λιβύη, γιατί έχει κάνει τεράστια βήματα. Σωστό είναι αυτό, αν δείτε και τι γίνεται στην όμορφη χώρα την Αίγυπτο. Είναι άδικη αυτή η εικόνα. Γιατί φυσικά πάντα ξέρετε ότι τα διεθνή ΜΜΕ εστιάζουν στα άσχημα, στα προβλήματα. Φυσικά υπάρχουν και σημεία επιτυχίας, αλλά δεν εστιάζουν σε αυτά. Είπα λοιπόν στους ε, συνομιλητές μου ότι είναι προς το συμφέρον τους να ρυθμίσουν το διπλωματικό θέμα με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ελπίζω ότι αυτό θα ανοίξει το δρόμο για πιο στενή συνεργασία με το δικαστήριο. Επίσης, είπα, όπως είπε και το δικαστήριο, ότι θα ήταν πολύ σημαντικό η Λιβύη να δικάσει αυτούς τους υψηλά ιστάμενους του καθεστώτος Καντάφη ε, και τον Σαϊφ και έτσι θα αποκτήσει αξιοπιστία θα είναι σημαντικό. Επίσης, είναι σημαντικό να υπάρξει και διεθνή υποστήριξη για όποιε τι διαδικασίες και από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ε, θα τη δώσει αξιοπιστία. Και όλοι οι συνομιλητές μου συμφώνησαν με αυτό. Να σας πω επίσης ότι είναι πολύ σημαντική δουλειά που μπορεί να κάνει το δικαστήριο, ούτως ώστε να προχωρήσουν οι δικαστικές έρευνες για τους βιασμούς ε, και τα εγκλήματα γενοκτονίας ε, εναντίον ανδρών και γυναικών το Μιζουράτ και αλλού στη Λιβύη. Καταλαβαίνετε τις τεράστιες ευαισθησίες που έχουν, έχει αυτός ο συντηρητικός λαός πρέπει να το λάβει υπόψη στη διεθνή κοινότητα. Αλλά υπάρχει και υποστήριξη από το λιβικό λαό α, να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Ε, πολλοί έδωσαν καταθέσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, προσέφηκαν ως μάρτυρες. Ε, θέλω να σας ρωτήσω τώρα, τι κάνει το δικαστήριό σας, μιλήσατε για την υπόθεση του Ζανούση, που είναι κάτοικος Μαυριτανίας ε, που είναι αυτή τη στιγμή μάλλον στη Μαυριτανία, συγγνώμη, θα πρέπει να εκδοθεί ε, στο Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Αλλά και ο Μουσακούσα που συνεργάστηκε με τι Ευρωπαϊκέ Υπηρεσίε Πληροφοριών για θέματα όπως βασανιστήρια που υπέστησαν άνθρωποι κατά τη διάρκεια των μυστικών πτήσεων και των απαγωγών τη CIA. Ο Μουσακούσα, από ό,τι ξέρω, είναι στη Σαουδική Αραβία. Γιατί δεν ασκεί κανένα πίεση στην Σαουδική Αραβία να εκδώσει τον, τον κύριο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα. βάζω ένα σημείωμα ε, που θα αναφέρει όλα αυτά τα τελευταία απορίσματα τα οποία προέκυψαν από τις τελευταίες μου επαφές και θα τα μοιράσω σε όλους σας. Ευχαριστώ κύριε Γκόμες για αυτή την παρουσίαση. Τις απόψεις σας, πληροφορίες. Και τώρα παρακαλώ τον κύριο Σαλαφράγκα να πάρει το λόγο. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να καλωσορίσω του εκπροσώπου του Εθνού Ποινικού Δικαστηρίου. Το Κοινοβούλιο μα έχει σταθερή δεσμεύση με τι δράσει του Δικαστηρίου τόσο όσον αφορά την πολιτική του στήριξη όσο και στην εφαρμογή των θέσεών του στις συμφωνίες που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες. Σε αυτή την περίπτωση η υποστήριξη αυτών που έχουν συλληφθεί στη Λιβύη είναι μια από τις προτεραιότητες για μας. Είναι δύσκολο νομίζω να αγνοήσει την κατάσταση στη Λιβύη αυτή τη στιγμή. Ξέρετε όλοι ότι έχουμε δεσμευτεί για την υποστήριξη της μεταβατικής διαδικασίας. Πρόσφατα επισκεφθήκαμε και τον ε, αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση στη Λιβύη και όπω ο κ. Κόμε, θα πρέπει βεβαίω να συμμεθεί η πρόεδρο όσον αφορά την θεσμική σταθερότητα και τον εκδημοκρατισμό του κράτους. Όλοι γνωρίζουμε τις διαδικασίες που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στη χώρα και θα πρέπει να κάνουμε μια επαλήθευση της δικαιοδοσίας σε σχέση με τις πράξεις των λιβικών αρχών. Θεωρούμε ότι η χώρα μετά από την εποχή του Σενταματάρχη Κατάφη έχει επιστρέψει σε μια φάση που όλα θα πρέπει να γίνουν από την αρχή. Όχι μόνο βέβαια για θέματα ασφάλειας όπου έχουμε 4.000 χιλιόμετρα συνόρων χερσαίων και 2.000 χιλιόμετρα θαλασσίων, θα πρέπει επίσης να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να υπάρχει μια ε, αστυνομία που θα ανταποκρίνεται όσο περισσότερο στις επιταγές του διεθνούς δικαίου. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω ποια είναι η εντύπωση που έχετε για αυτή τη διαδικασία η οποία εξάγεται σχέση με αυτά τα τρία άτομα και ποια είναι η κατάσταση των δικαστικών αρχών της χώρας ώστε να μπορεί να εφαρμόσει όλα αυτά τα πράγματα. Και τι γίνεται με την κατάσταση ασφαλείας στην οποία βρισκόνται οι κρατούμενοι. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε κάτι σε σχέση με την μεταχείριση γιατί έγινε λόγος για και κακομεταχείριση και για βασανισμούς, το αναφέρατε εσείς προηγουμένως. Τι γίνεται λοιπόν με αυτά τα άτομα τα οποία ήταν του καθεστώτος Καντάφη. Αξιτάζεται και αυτές τις ε, υποθέσεις ή αφορούν μόνο την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτά ήθελα να μάθω. Η κυρία Γκόμες αναφέρθηκε στην περίπτωση Σαουδικής Αραβίας. Εγώ πρώτα θα ήθελα να μάθω ποιες είναι οι δράσεις του συμβουλιου ασφαλειας αυτα ηθελα να μαθω η κυρια γκομες αναφερθηκε στην περιπτωση Αδική Αραβία. εγω πρωτα θα ηθελα να μαθω ποιε ειναι οι δράσει του Διεθνού δικαστηριου που αφορούν την περίπτωση του πρόεδρου της Συρίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σαλφράγκα. Η κυρία Λόχπελης τώρα, πρόεδρος της Υποεπιτροπής των Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τους προσκεκλισμένους μας για τις εκθέσεις. Από τις 3 μέχρι τις 5 Ιουνίου ήμουν στην Τρίπολη της Λιβύης και ε, μετά την αποχώρησή μου μόνο έλαβε χώρο το περιστατικό της ε, σύλληψης των συνεργατών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Οπότε σε αυτό δεν έχω τίποτα να πω, αλλά είχαμε συζητήσει ε, και με το μεταβατικό συμβούλιο, με τον πρόεδρο δηλαδή, του μεταβατικού συμβούλιο, με τον ε, υφυπουργό, τον αρμόδιο για, στη μεταβατική κυβέρνηση για τη δικαιοσύνη και με άλλους ε, εκπροσώπους μεταβατικής κυβέρνησης με κύριο ερώτημα αν προτίθεται να κυρώσει το καταστατικό του Εθνούς Ποινικού Δικαστηρίου η Λιβύη ε, η οποία πήρε σαν απάντηση ότι δεν βλέπουν γιατί τόσο γρήγορα και τόσο πρόημα και τόσο πιεστικά τους στήθησε αυτό το ζήτημα. Επίσης, ε, ως προς το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, σημειώνεται από πλευράς της Λιβύης ότι χαιρετίζεται το καταστατικό αυτό, αλλά ταυτόχρονα δεν γίνονται δεκτέοι οι πενιγμοί ότι ο Σαΐφ Αλισλάμ ενδέχεται να μην λάβει δίκη σε επίπεδο ισότιμο με αυτό των διεθνών, της διεθνούς κοινότητας, εάν δικαστεί μέσα στην Λιβύη. Σε αυτό επιμένουν πάρα πολύ. Και γι' αυτό θα ήθελα να ερωτήσω, εάν κάποιος δικαστή ε, με το λιβικό δίκαιο ενώπιον ε, λιβικού δικαστηρίου υπηκρέμεται ακόμη και η ποινή του θανάτου. Άρα σε αυτό προφανώς υπάρχει διαφορά και ασυμβατότητα με το καταστατικό του Εθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είχε να κάνει με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ήταν ότι όπως μου είπαν ναι δέχονται, θα θέλαν να συνεργάζονται με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αλλά δεν μπορούν να έχουν τον έλεγχο πάνω στους ε, κρατουμένους που έχει στα χέρια της ε, η πολιτοφυλακή και ως εκ τούτου δεν μπορούν να προχωρήσουν στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις αυτές. Άρα λοιπόν και από ό,τι λένε θα προσπαθήσουμε με βάση και τις εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν ελπίζουν με τις ε, βέλτιστες ε, προδιαγραφές να ανακτήσουν τον έλεγχο στις ε, πολιτοφυλακές αυτές. Ξέρω ότι είναι δύσκολο βέβαια να τοποθετηθεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στο θέμα αυτό, αλλά θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση και αν αλλάξει μπορεί αυτές οι πολιτοφυλακές να δεχθούν να παραδώσουν τους κρατουμένους τους. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Ντόρφερ που είναι και εισηγητής για το Διεθνές Δικαστήριο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Και ευχαριστώ πολύ για την διεξοδική ε, παρουσίαση των θέσεών σας, την κυρία Γκόμες, την κυρία Λόχμπιλερ επίσης, η οποία όπως είδατε είναι πολύ, επίσης, όπως είναι πολύ με την κατάσταση στη Λιβύη. Θα ήθελα να πω ότι είναι εμφανές ότι η διεθνής απήχηση που θα έχει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από το πώς θα επιληθεί το ζήτημα της Λιβύης και πώς οι ε, αρχές της Λιβύης ή αυτοί που έχουν την ευθύνη της ε, ε, καθοδήγηση της χώρας θα συνεργαστούν, εάν συνεργαστούν με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Γιατί από αυτό θα κριθεί και το πώ θα διαμορφωθούν σαφεί δομέ, δικαστικέ δομέ στη Λιβύη. Ξέρουμε, όπως ανέφερε και η κυρία Λόχ Μπίτλερ, σε πιο μεγάλο βαθμό οι ε, μουσουλμάνοι αδελφοί όταν ήρθαν στο ε, Μόναχο ε, ξέδωσαν τρόπον την Α, πήγαν σε δισκοτέκ, έκαναν τη μεγάλη ζωή, εν πάση περιπτώσει ξέφυγαν από αυτό το οποίο θεωρητικά παρουσιάζουν ως τρόπο ζωής. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ή καλύτερα να παραλείψει κάποια πράξη η οποία θα είχε ενδεχομένως ε, ε, βλαπτικό αποτέλεσμα, δηλαδή σχόλια τα οποία ίσως δημιουργούν δυσκολότερες ε, συνθήκες, είναι αντιπαραγωγικά δηλαδή ως προς τη σχέση σας με την ηγεσία της Λιβύης. Γιατί είναι σημαντικό βέβαια να τοποθετούμε θα ξεκάθαρα, αλλά από την άλλη έχει επαφεθεί λίγο πολύ στα χέρια της κυρίας Κάθη Άστον η διαμόρφωση μιας κοινή θέση από πλευράς των Υπουργών των Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ίσως κάποια κράτη έχουν πιο άμεση εμπλοκή και θα ήθελα να έχουν πιο σοφή τοποθέτηση. Επίσης, στα Ηνωμένα Έθνη έχει λίγο πολύ ε, δοθεί η επίσημη τοποθέτηση με το ανακοινωθέν τύπου ότι θα πρέπει το Διεθνές Ποινικό Δικαστηρίο να δράσει ανεξάρτητα και να ε, προχωρήσει όπως επιλέγει. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν νομίζετε ότι έχετε επαρκή, επαρκές ειδικό βάρος για το καθήκον το οποίο αναλαμβάνετε και αν χρειάζεται κάποια άλλη βοήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κράσιλ Τέρφερ και τώρα η κυρία ε, Μπραντνερ. Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και τους προσκεκλημένους μας. Θα ήθελα να ρωτήσω, μια και αναφερθήκατε στην ε, προετοιμασία των ε, δικών από πλευράς των Λιβύων, συλλογή αποδεκτικών στοιχείων κτλ. Δουλειά που έχετε ήδη κάνει εσείς και εσείς έχετε μαζέψει αποδεκτικά στοιχεία. Εσείς έχετε στοιχειοθετήσει την υπόθεσή σας. Ε, ρωτώ λοιπόν σε ποιο βαθμό υπάρχει συνεργασία, εάν υπάρχει, στη συλλογή των αποδείξεων. Το ρωτώ αυτό διότι ίσως, ίσως όχι άμεσα βέβαια, αλλά σε μεσοπρόθεσμη πρόπτικη μέσα σε ένα χρόνο φερειπίνησης να υπάρχει δυνατότητα να διεξαχθούν πράγματι δίκες αυτές σε ικανοποιητικό επίπεδο μέσα στη Λιβύη. Πώς θα το χειριστείτε αυτό. Και αυτό βέβαια εντάσσεται και στη γενικότερη συζήτηση για το κατά πόσον είναι σε θέση η χώρα να χειριστεί το θέμα των αποδείξεων αλλά και άλλα ζητήματα όπου ίσως να μην έχετε ξεκινήσει στις μεγάλες δίκες, αλλά στοιχεία έχετε στα χέρια σας. Πληροφορίες έχετε. Τι θα τις κάνετε λοιπόν αυτές τις πληροφορίες, έστω και αν δεν μπορείτε να στραφείτε δικαστικά κατά των ανθρώπων αυτών, θα τις ε, διαβιβάσετε σε κάποιον επιτροπή συμφιλίωσης, μεταβατικό συμβούλιο Μην ξεχνάμε ότι χρειάζεται κάποια στιγμή οι άνθρωποι, η, η Λιβύη να έρθει αντιμέτωπη με, το, με την ιστορία της και να ξεκινήσει μια διαδικασία συμφιλίωσης. Πώς θα το χειρίσετε λοιπόν αυτό. Έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις όπου υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, αλλά ίσως ε, δεν θέλετε να προσαγάγετε, δεν μπορείτε να προσαγάγετε κάποιους. Και κάτι ακόμη σχετικό με τη Σαουδική Αραβία που πιστεύω θα πρέπει να τεθεί. Ε, διότι πρέπει να πούμε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δίνει την εντύπωση ή τρέφεται η εντύπωση για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ότι δεν αντιμετωπίζει τους πάντες με τον ίδιο τρόπο. Στο θέμα λοιπόν της Σαουδικής Αραβίας πώς και τι ακούτε, τι σκοπεύετε να κάνετε, πιστεύετε ότι πρέπει να δώσετε περισσότερη προσοχή στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Άλλες δύο παρεμβάσεις, ο κύριος Μάιερ από την ΚΟΕ, Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Την εκπρόσωπο του Διεθνούς Δικαστηρίου, καταρχήν να εκφράσω την αλληλεγγύη της ομάδας μου με τους τέσσερις εκπροσώπους του Δικαστηρίου που απήχθησαν ακριβώς μιας κυβέρνησης η οποία δεν κυβερνά δεν κυβερνά τη Λιβύη αποτέλεσμα μιας ε, στρατιωτικής επέμβασης που ήταν ε, καταστροφική, δηλαδή αυτή του ΝΑΤΟ. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ήταν καταστροφική η επέμβαση του ΝΑΤΟ. Ήταν καταστροφική. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να συνεχίσω χωρίς να με διακόπτουν. Ε, ήταν λοιπόν καταστροφική επειδή δεν τήρησαν, δεν εφάρμοσαν μάλλον την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν είχαμε την ζώνη αποκλεισμού για την προστασία του πληθυσμού. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Μετατράπηκαν στη αεροπορία της αντιπολίτευσης του Μεταβατικού Συμβουλίου. Αυτό ήταν και από αυτή την κατάσταση προκύπτουν όλα αυτά τα προβλήματα τώρα. Ο εκπρόσωπο της κυβέρνηση Μοχάμετ Αλσερέτσι είπε ότι οι τέσσερις εκπρόσωποι, εντάξει αυτόν και ένα Ισπανό, οι τέσσερις λοιπόν εκπρόσωποι του Διεθνού Δικαστηρίου θα απελευθερωθούν όταν παράσχουν πληροφορίες για το που βρίσκεται ο Ισμάδε Σαφίν, ο οποίος είναι ένας από τους βοηθούς του γιου του Κατάφη. Αυτό είναι μια απαγωγή λοιπόν με στόχο την παροχή πληροφοριών απαγωγή, ξεκάθαρα. Γι' αυτό σας παρακολουθώ ή μην μιλάτε για συλλήψεις. Πρόκειται για απαγωγή. Αν τους δώσουν τις πληροφορίες από το Εθνές ε, Επιτικό Δικαστήριο, τότε αφήνονται ελεύθεροι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Απολύτως απαράδεκτο. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το χαοτικό πλαίσιο όπου έχουμε πολιτοφυλάκες, όπου έχουμε διάφορες φυλές, φιλάρχους κλπ. Έχουμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο χιλιάδες συλλήψεις και κρατούμενους που δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Και βέβαια το Διεθνές Δικαστήριο θα έχει όλη την υποστήριξή μας, κάθε υποστήριξη από εμά, ώστε να οδηγεί στο δικαστήριο όλους τους υπεύθυνους και από το καθεστώς Καντάφη και από το καθεστώς που τον διαδέχτηκε. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνήσουμε τι γίνεται και με την βάρβαρη εκτέλεση του δικτάτορα Καντάφη, γιατί οι εικόνες που είδαμε δεν θα πρέπει να μείνουν ατιμόρυτες. Εκτός και αν φαίνεται αυτό στον νόμο του αίματος, αποδεχόμαστε ότι είναι τμήμα αυτού του πολιτισμού. Βεβαίως θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνε και στο καθεστώ Καντάφη αλλά και στο μεταβατικό καθεστώ. Νομίζω είναι εξίσου σημαντικό. Οπότε οι πληροφορίε που μα έδωσαν για αυτέ τι 26.000 επιδρομέ, αεροπορικέ επιδρομέ, οι 26 αυτέ χιλιάδες αεροπορικέ επιδρομέ προκάλεσαν πολλά αθώα θύματα για το οποίο θα πρέπει κάποιο και γι' αυτά να αναλάβει ευθύνη. Δεν θα πρέπει λοιπόν να παραβλέψουμε ευθύνες, είτε πρόκειται για πιλότους βαμβαδιστικών του ΝΑΤΟ, είτε για αξιωματούχους ή αξιωματικούς του στρατού του Καντάφη, είτε για εκπροσώπους της ε, ΑΛΚΑΙΔΑ. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ έχετε κάθε υποστήριξη από εμάς, ώστε να κάνετε τη δουλειά σας και να θέσουμε ένα τέλος σε αυτή την απαράδεκτη απαγωγή αυτό των υπαλλήλων. Θα πρέπει λοιπόν ως Κοινοβούλιο να απαιτήσουμε την ανεφόρον απελευθέρωση των εκπροσώπων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ευχαριστώ πολύ. I Στο κύριε Μάιερ, ο κύριος Κυρίλοφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια άλλη διάσταση θέλω να θέσω. Για τον Σαΐφ Αλισλάμ θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποφασιστικοί και θα πρέπει να έχουμε μια κοινή θέση. Γιατί δεν μπορούμε να φτάσουμε σε κοινή θέση. Και τα θέτω και στον εαυτό μου ερωτήματα σε σχέση με αυτό. Καταρχάς, για κάποιο χρονικό διάστημα ο Σαΐφ ήταν ο μεταρρυθμιστής του καθεστώτος. Ε, περιφερόταν σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, είχε συναντήσεις με υψηλά ιστάμενους, ε, υπέβαλε κάποιες πρωτοβουλίες και από ό,τι ξέρω είχε καλή υποδοχή η προσπάθειά του. Είχε και πολύ σημαντικές πληροφορίες μέσα στην κατοχή του. Ίσως γι' αυτό δεν ασκούμε μεγάλη πίεση. Δεύτερον, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη Βουλγαρία είχαμε μια, αυτή την ιστορία με το προσωπικό, α, της νοσοκόμες και τα λοιπά, που τις είχα, είχαν καταδικαστεί σε θάνατο τρεις φορές. Αλλά αυτός ε, έπαιξε διαφορετικό ρόλο, μεταρρυθμιστικό. Και τώρα μάλιστα υψηλά στάμενη πολιτική ε, στη Λιβύη συμμετείχαν στην κακομεταχείριση του ιατρικού μας προσωπικού. Ε, τις κατηγόρησαν αυτές τις νοσοκόμες ότι σκότωναν παιδιά. Ε, και γιατί τα λέω τώρα όλα αυτά. Γιατί θέλουμε να πάει ενώπιον του δικαστηρίου ο Σαϊθ Ισλάμ. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το πετύχουμε αυτό. Αυτό, αυτό θα έχει και επίπτωση για ορισμένους πολιτικούς σήμερα στην κυβέρνηση. Ε, θα πρέπει όμως εμείς να το πετύχουμε αυτό και να ασκήσουμε πίεση για να το πετύχουμε. Έχετε την αίσθηση και εσείς ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ως Γιατί εγώ έχω αυτή την εντύπωση. Ευχαριστώ κύριε Κυρίλο. Πολύ σημαντικά αυτά τα σχόλια. Θα δώσω τώρα το λόγο στους προσκεκλημένους μας για να προσπαθήσουν να απαντήσουν σε ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών επί των διαφόρων σημείων που ακούστηκαν. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Και δεν θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τις πολύ καλές ε, προτάσεις και την υποστήριξη από τους ε, συναδέλφους που είχαν πρόσφατα επισκεφθεί την Λιβύη. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η υποστήριξη που μας προσφέρετε για τη δουλειά μα. Θα προσπαθήσω να δώσω τι απαντήσει Αν τυχόν λησμονήσω καμιά ερώτηση, συγχωρήστε με. Αναφερθήκατε στον Παγκραντή, τον Μουσακούσα, Κάμπας και άλλα πρόσωπα τα οποία θα έπρεπε ίσως να διερευνήσουμε. Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε τη συλλογή των στοιχείων, συνεχίζουμε την ε, έρευνα. Είμαστε ποινικό δικαστήριο και άρα θα πρέπει να συνδέσουμε ε, χωρίς ε, την παραμικρή αμφιβολία πρόσωπο με αδίκημα. Είμαστε ποινικό δικαστήριο και δεν ξεκινήσαμε με την ε, πρόθεση ότι θα εκδικάσουμε κάθε έναν, κάθε μία υπόθεση θα δικάσουμε κάθε έναν ύποπτο. Ε, κοιτάμε τα πιο σοβαρά αδικήματα Κοιτάμε αυτούς που είναι οι πλέον υπέτη για τα πιο σοβαρά αδικήματα. Αλλά για τα θέματα τα οποία επισημαίνεται πρέπει να σας πω ότι συνεχίσουμε τις ανακρίσεις, ε, την έρευνα και θα συνεχίσουμε όσο χρειάζεται. Όπως είπατε και εσείς, είναι περιορισμένος ο προπολογισμός μας. Και αυτό επηρεάζει επίσης το πόσο γρήγορα μπορούμε να κινηθούμε αυτό επηρεάζει επίσης το ε, κατά πόσον μπορεί κάπου να προσκρούσουν ε, οι διαδικασίες αυτές οι ερευνητικές και να χρειαστεί να σταματήσουμε, να διακόψουμε για λίγο. Για το κατά πόσον μπορούμε να περιμένουμε από τους ε, Λιβύους την διεξαγωγή μιας αντίστοιχης δίκης της δίκης. Αυτό εξαρτάται από το ρόλο των δικαστηρίων και του δικαστηρίου του δικού μα. Εμεί δεν εξετάζουμε πάλι ολόκληρο το δικαστικό σύστημα στη Λιβύη. Κοιτάμε πολύ μεγάλη προσοχή και οι δικαστέ μα θα εξετάσουν πολύ μεγάλη προσοχή. Εάν όντω ε, οι διαδικασίε που βλέπονται οι δικαστικέ ε, είναι για τα ισοδύναμα εγκλήματα ισοδύναμες. Δεν θα κάνουμε εμεί επισκόπηση όλου του συστήματο, τη δικαίωση του κεσικού συστήματο τη Λιβύη. Αυτό δεν είναι δική μα δουλειά. Πολύ συγκεκριμένε περιστάσει εξετάζουμε μόνο και βέβαια και το ποσοστό της λεγόμενης δίκαιης δίκης εφόσον τηρείται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο πάλι θα ε, συνυπολογιστεί. Ο κίνδυνος να επιβληθεί θανατική πηγινή. Κοιτάξτε, εδώ δεν έχουμε δει άλλη αντίστοιχη περίπτωση στο παρελθόν. Είναι άνευ προηγουμένου δηλαδή οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε και άρα θα πρέπει να βρούμε λύσεις δεν λέγεται πουθενά στο καταστατικό ότι η συμπληρωματικότητα δεν ισχύει εφόσον υπάρχει κίνδυνος για πιο αυστηρή ποινή στην ίδια τη χώρα από ό,τι θα μπορούσε να επιβάλλει το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Ξέρουμε ότι αυτό αφορά δύο συγκεκριμένε περιπτώσει, αλλά εν πάση ο συνάδελφο μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία. Πάντω δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη στο καταστατικό μα. υποστηρικτές του Καντάφη. Κοιτάξτε, η εντολή που μας έδωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας είχε να κάνει με τα εγκλήματα μέχρι τις 15 Απριλίου του 2011 και ήταν ξεκάθαρο ότι κοιτάμε, ε, ε, εξετάζουμε δικήματα από οποιαδήποτε πλευρά, όχι μόνο της μίας πλευράς, αλλά πάλι, παραλαμβάνω, όχι όλα τα αδικήματα ανεξαιρέτως. Κοιτάμε ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος και τη σοβαρότητα της επαιτειότητας. Πάντα κοιτάμε τα πιο σοβαρά αδικήματα και κάνουμε στο δυνατόν πιο αδέκαστη και ουδέτερη ε, έρευνα. Και αυτό φυσικά στρέφεται κατά των πάντων. Εάν υπάρχουν τώρα αδικήματα εις βάρος των ε, κρατουμένων, δηλαδή αν ε, υπάρχουν αιτιάσει για τις αρχές ασφαλείας, δεν αποκλείεται να συνεχίσουμε την ε, διαρεύνηση, εφόσον συλλέξουμε αρκετά στοιχεία. Αλλά πάντως και τα, και τα σχετικά με, με τη γενετήσια ελευθερία και το, το φύλλο περισσότερο θα τα εξετάσουμε περαιτέρω. για την ε, κατάσταση στην οποία αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι. Κοιτάξτε, κρατούμενοι είναι. Δεν έχουμε καμιά ένδειξη ότι τους κακομεταχειρίζονται. Έχουν τύχει καλή μεταχείριση από ό,τι γνωρίζουμε. Έχουμε μια συντονισμένη προσπάθεια βέβαια. Η κυρία Άστον ασφαλώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στην υπόθεση αυτή. Είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια του συντονισμού. Το Συμβούλιο Ασφαλείας έκανε την Παρασκευή δήλωση όπου επισημαίνει σοβαρές ανησυχίες για την κράτηση και όπου καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές της Λιβύης να συνεργαστούν για την ταχεία αποφυλάκηση, απελευθέρωση καλύτερα των κρατουμένων. Φυσικά περιμένουμε την υποστήριξη, θέλουμε την υποστήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν έχουμε ενδείξει ότι θα συμβεί κάτι διαφορετικό στο εκείς μέλλον. Αλλά πάντως ήταν σημαντική αυτή η υποστήριξη μας προσέφερε με τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η περίπτωση να έχουν διαπραχθεί αδικήματα στη Συρία, τη Σαουδική Αραβία ή αλλαχού. Κοιτάξτε, το, καθεστώ, το καταστατικό μας, το καταστατικό της Ρώμης ε, αναφέρεται στην δικαιοδοσία μας ξεκάθαρα με βάση το κεφάλαιο 7 του καταστατικού των Αθηνών με την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας ορίστε ξεκάθαρα η δικαιοδοσία που έχουμε. Ε, συγκεκριμένα για τη Συρία, τη Σαουδική Αραβία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διότι τους άλλους δεν είναι και συμβαλόμενα μέρη. Επομένως, αν έχουν διαπραχθεί σχετικά δικήματα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα διαβάζουμε σε εφημερίδες. Γιατί ποτέ περισσότερο. Τα άλλα είναι στο χέρι του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το ίδιο και για την οικουμενικότητα των ανθρωπινών δικαιωμάτων που αναφέρεται. Γιατί εδώ ουσιαστικά έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα. Ένα σύστημα για τα συμβαλόμενα μέρη. Ένα βασικό εργαλείο δηλαδή για να σταματήσουν τα μαζικά εγκλήματα ε, και να κληθούν να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για αυτά, οι υπέτειοι για αυτά. Και το άλλο το οποίο είναι στα χέρια του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ε, όσο πιο πολλά κράτη δηλαδή ε, ενσωματωθούν ε, στην σύμβαση, στο διεθνέ σύστημα, τόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι το σύστημα της λογοδοσίας. Επίσης, στο να δίνουμε πληροφορίες με, σε κράτη-μέλη. Δεν προβλέπεται τίποτα από το 9310 ώστε να δίνουμε σε κράτη, -μέλη, σε κράτη άλλα, σε τρίτα κράτη στοιχεία στη Λιβύη εν προκειμένου. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μέχρι τώρα έχει πάει καλά η συνεργασία, αλλά επειδή πρόκειται για μια δικαστική διαδικασία, εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να δώσουμε δηλαδή συμβουλές ε, δικαιοδοτικού χαρακτήρα, γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να δικάσουμε εμείς τις υποθέσεις. Και πάντα διατηρούμε μια κάποια απόσταση με γενικόλογες εκφράσεις. Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι οι διαδικασίες όπως θα έπρεπε κτλ. Αλλά τίποτε περισσότερο. Πάντως και στη συλλογή των αποδείξεων και σε άλλα ε, σχετικά θέματα δεν είδαμε προβλήματα, δεν είδαμε δυσκολίες και δεν περιμένουμε στο μέλλον. Για το αν υπάρχουν πιέσεις να μην προσαχθεί ο Σαΐφ Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί η σημασία του να συνεργάζονται τα κράτη με το δικαστήριο και βέβαια ε, αυτό έχει να κάνει και με την ε, ένσταση παραδεκτού. Πρέπει να το δεχθούμε αυτό και πρέπει να συνεργαστούν και οι ε, αρχές της χώρας μέσα στο καταστατικό ώστε να εξασφαλιστεί η γενικότερη λογοδοσία είτε πρόκειται για εθνικές ε, διαδικασίες δεν πρόκειται για τις ε, αποφάσεις των, δικα, των δικαστών του Διεθνούς αν Θέλει κάτι να προσθέσει και συνάδελφος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω. Θέλω να σταθώ σε μερικά σημεία που ακούστηκαν. Εγώ ασχολούμαι, ε, είμαι στην Χάγη, ε, στην ερευνητική ομάδα. Αρχίσαμε να δουλεύουμε τον Νοέμβριο για αυτό το θέμα. Είχαμε καλή συνεργασία με τις Λιβικές Αρχές. Ε, στην προσπάθεια διερεύνησης των υποθέσεων. Μας έδωσαν δηλαδή πολλά στοιχεία, πολλές αποδεικτικές στοιχεία, πολλά αποδεικτικά στοιχεία και εκείνοι συνέλεξαν μάλιστα τέτοια, τέτοιες αποδείξεις. Ο Μαχμούδ Μπαγντάτι, ο πρωθυπουργός, ο Αλ Ισλάμ κτλ. Ε, έφυγαν και άφησαν τα γραφεία του άθικτα. Όλα λοιπόν τα έγγραφα υπήρχαν και τα είχε στην κατοχή, τα έχει στην κατοχή το Εθνικό Μεταβατικό Συμβούλιο. Ε, υπήρχαν χιλιάδες χιλιάδων υποκλοπές ε, τελεφωνικές κτλ. Ε, τον Απρίλιο λοιπόν ε, ήμουνα με το Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος εξήγησε τι στοιχεία είχε. Έχουμε κάποια, αποδείξεις μας εν μέρη συμπίπτουν, έχουμε και παραπάνω. Ή μάλλον εκείνοι είχαν παραπάνω οι λιβικές αρχές. Κάναν σοβαρές λοιπόν ανακρίσεις, σοβαρές έρευνες αλλά όπως είπε και οι συνάδελφοι, οι δικαστές θα πάρουν τελική απόφαση. Δεν είναι εύκολο να πούμε εμείς πώς θα αντιδράσουν οι δικαστές. Μπορεί να αποφασίσουν να κάνουν προφορικές διαδικασίες, ε, όπως έχει ζητηθεί, αλλά εξετάζεται ακόμα το αίτημα. Απλώ θα βάλουν χρονοδιάγραμμα στις ε, διαδικασίες. Θα, δεν θα δώσουν ένα πλήρε πράσινο φω, θα πούν στι λιβικέ αρχές, ξαναελάτε, α πούμε, και ε, σε επαφή μαζί μα για να δούμε τι θα γίνει. Ε, όλη αυτή η δικασία για του Λίβιου είναι πολύ σημαντική. Όταν συναντηθήκαμε με την Τρίπολη, με το Γενικό Εισαγγελέα, ε, προστάτευσε ας πούμε, την περιοχή του ας πούμε, και το, τα στοιχεία που είχε κτλ. Είπε ότι είσαστε απ' έξω, α πούμε. Είναι σημαντικέ οι ανακρίσει μου κτλ. Ίσως ε, το 85% από αυτά που κάνει ε, θα μπορούσαν να δημοσιοποιηθούν. έχει υποβληθεί μία, ένα αίτημα για την έγκριση όχι του παραδεκτού. Επομένως λοιπόν, έχουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα, προσπαθούμε να δούμε τι κάνουν όλοι οι φορείς και πώς μπορεί να συνεισφέρει το ποινικό δικαστήριο. Για το θέμα της θανατικής ποινής θα ξέρετε ότι έγινε μεγάλη συζήτηση στη Ρώμη και υπήρχαν ακρές απόψεις και στις δύο πλευρές του φάσματος. Από ό,τι ξέρω, υπάρχει και μια διάταξη στο καταστατικό που λέει ότι το καταστατικό δεν απαιτεί από τα κράτη να αλλάξουν τη θέση τους σε ό,τι αφορά τη θανατική ποινή. Α, αλλά συμφωνώ ότι ίσως αυτό είναι ένα θέμα που οι δικαστές του δικαστηρίου θέλουν να λάβουν υπόψη ε, και είναι ένα καινούριο θέμα, ένα καινοφανές θέμα. Ε, η Λίβη στο Συμβούλιο Ασφαλείας έκανε το Μάιο μια πολύ σημαντική παρέμβαση, στις 16 Μαΐου συγκεκριμένα. Ο εκπρόσωπος ε, των Λίβιων είπαν ότι θεωρούσαν ότι είναι σημαντικό να υπάρξει λογοδοσία για κάθε θύμα της Λιβύης, α, όποιος και ήταν ο Αυτό θα πρέπει να, αυτό θα πρέπει να σημαίνει ίσως το να υπάρξει μια ιεράρχηση Τη σημασία των υποθέσεων. Ε, ίσως ε, τα εγκλήματα πούμε, του Γκαντάφη είναι πιο ψηλά στην ατζέντα, αλλά γενικά θα υπάρξει μια ιεράρχηση και... Και εμείς κάνουμε ερωτήσεις του τύπου ε, τι επιπτώσεις θα έχει αν ας πούμε διερευνήσετε τυχη υπόθεση και όχι την ψή προσπαθούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε κι εμείς, εν πάση περιπτώσει, την όλη διαδικασία. Ο κύριος Κυρίλοφ, δεν με σχολιάσατε το ερώτημά μου, συγγνώμη. Το οποίο ήταν, αν πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιοι, είτε εδώ είτε στη Λιβύη, που δεν επιθυμούν να προσαχθεί ο Σαΐφ Αλισλάμ στο δικαστήριο και πιστεύετε ότι χρειάζεται πολιτική πίεση για να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Συγγνώμη. Προσπάθησα να το απαντήσω διπλωματικά. Ίσως ήμουν υπερβολικά διπλωματική. Ναι, ναι, ήμουν πολύ διπλωματική στην απάντησή μου. Η πίεση θα πρέπει να υπάρχει σε συνεργασία με το δικαστήριο. Να λογοδοτήσει ο ΣΑΙΦ. Ε, είτε στο δικαστήριο είτε στις εθνικές αρχές. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, θα αποφασιστεί. Πάντα υπάρχουν άτομα που δεν θέλουν κάποιοι ψηλά ηθήνοντες, ας πούμε, να λογοδοτήσουν. Όλοι μας θα πρέπει να πιέζουμε για να υπάρξει λογοδοσία. Δεν χρειάζεται ε, να αποφασίσει δεν και καλά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αν αποφασίσουν δικαστές ότι μπορούν να το κάνουν οι λιβικές ε, δικαστικές αρχές, μπορεί να γίνει και έτσι. Ένα σχόλιο από την κυρία Γκόμε. Από τις επαφές που είχα αυτό το Σαββατοκύριακο με του Λίβιου, προκύπτει ότι υπάρχει αντίληψη ότι κάποιοι θέλουν να αθωωθεί, να απαλλαγεί ο Σαΐφ, ε, να μην προσαχθεί καν σε δίκη και μάλιστα να τον αφήσουν να συνομωτήσει εναντίον του σημερινού καθεστώτος. Ακριβώς γι' αυτό ε, υπάρχει αυτή η φοβερή παρεξήγηση και αυτή η προκατάληψη εναντίον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Η κοινή γνώμη το πιστεύει αυτό. Παρότι καταλαβαίνει ότι αυτό δημιουργεί μια άσχημη ας πούμε, εντύπωση για τη Λιβύη στο εξωτερικό. Και θέλουν να συνεργαστούν με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτό είναι ο λόγο. Υπάρχει αυτή η παρεξήγηση από πλευρά Λιβύων. πιστεύουν, αυτό πιστεύουν. Και έτσι δικαιολογούν ας πούμε, και αυτή την κράτηση ή την απαγωγή ας πούμε, του το προσωπικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ε, για τους υποστηρικτές του Γκαντάφη, ε, ποια είναι η κατάστασή τους έτσι, από ανθρωπιστικής πλευράς. Θα μπορούσατε ίσως να απαντήσετε and Mr. Salafranca to make it clear the questions because it was not, uh, not clear. Ναι, ίσως να μην ήταν σαφή κάποια απάντηση η ερώτηση. ρώτησα κάτι και δεν απαντήθηκε σε σχέση με την εκτός δικαιοσύνης εκτέλεση του Κατάφη. Θα διερευνηθεί και αυτό. Κύριε Σαλαφράγκα, επίσης θέλετε να διευκρινίσετε είχαμε κατηγορίες σε σχέση με βασανιστήρια των υποστηρικτών του Καντάφη που είναι φυλακισμένοι. Δεν γνωρίζω τον αριθμό. Έχετε κάποια στοιχεία για τον αριθμό των κρατουμένων υποστηρικτών δηλαδή του Καντάφη. Έχετε το λόγο, κυρία Σουά Κόλμαν. Ναι, να απαντήσω σύντομα σε σχέση με τις δολοφονίες, με τη δολοφονία του κυρίου Καντάφη προσπάθησα και πάλι να απαντήσω διπλωματικά. Αλλά να πω ότι θα εξετάσουμε όλες τις δολοφονίες που αφορούν οποιοδήποτε. Και είπαμε προηγουμένως ότι πραγματικά μπορεί να είναι έγκλημα πολέμου η δολοφονία του Καντάφη και θα το εξετάσουμε. Θα πρέπει όμως να δούμε Ποιε υποθέσει θα πρέπει να εξετάσουμε υπό το φω της πληρωματικότητα, ποιε θα πρέπει να προωθηθούν, πώς θα συλλέξουμε τα στοιχεία κλπ. κλπ. Είναι κάτι για το οποίο έχουμε δικαιοδοσία και το οποίο ξέρουμε ότι αποτελεί έγκλημα σύμφωνα με την δικαιοδοσία μας και αυτό θα το εξετάσουμε. Το εξετάσουμε λοιπόν. Τώρα για τους κρατούμενους από τις δυνάμεις του Καντάφη. Έχουμε την έκθεση του Μάρτη 2012 που αναφέρει ότι έχουμε χιλιάδες κρατούμενους. Είχαμε ενδείξεις λοιπόν κακομεταχείρισης και ενδεχομένως βασανιστήριων. Αυτό για μας είναι προτεραιότητα και σε συναντήσεις με τους Λίβιους καταδείξαμε την ε, σημασία της απελευθέρωσης όπου πρέπει, την ε, σωστή δίκη, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων κλπ. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συλλέξουμε και άλλε πληροφορίε να κληρώσουμε η δικασία αυτή. Ναι, για την διερεύνηση της δολοφονίας του Καντάφη. Νομίζω ότι γι' αυτός ενδεχομένως δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα. Ίσως να υπάρξει και αρνητική αντίδραση. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι η δολοφονία του Καντάφη αποτελεί ένα κακό παράδειγμα όσον αφορά τη λογοδοσία και θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Για... για τη συνωμοσία που λέγαμε προηγουμένως. θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι δραστήριοι εκτός ε, Λιβύης και εμπλέκονται ακόμα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι ενδεχόμενη ευθύνη έχουν ακόμα για κλίματα υπό την εντολή μας βέβαια, στα πλαίσια της εντολής μας. Αν διαβάσετε τα ανακοινοθέντα τύπου θα δείτε ότι είναι ακόμα δραστήρια αυτοί, οι οικογένειές τους, και ίσως να υπάρχουν κάποια θέματα ασφάλειας που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με τους Λίβιους για το πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε μια τέτοια κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Σπακόλτμαν και κυρία Σέντς που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ε, παραφορά της δικαιοσύνης. Έχετε την υποστήριξή μας. Ευχαριστούμε. Okay, now we continue because we would like to... Συνεχίζουμε για να τελειώσουμε και έγκαιρα. Έχουμε την έκθεση για την εξωτερική πολιτική, για στρατηγική ψηφιακή ελευθερία στην εξωτερική πολιτική τη ΕΕ, κυρία Σάκη, η συγκίτρια, και τη ζητώ να παρουσιάσει την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε αυτό που θα κάνουμε σήμερα θα είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων βάσει του εγγράφου που με τους σκιώδεις αλλά και μαζί με, τους, με το κοινό online θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω κάποιες πρώτες εντυπώσεις πάνω στις οποίες θα βασίσω το προσχέδιο του, της επίσημης έκθεσης. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να συνεργαστούμε για να εκπονήσουμε την πρώτη στρατηγική ψηφιακή ελευθερία στην εξωτερική, εξωτερική πολιτική τη ΕΕ. Εδώ έχουμε κάποιες ε, επαστατικές εξελίξεις στον τομέα αυτό που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή, καθημερινή μας ζωή αλλά και την εξωτερική πολιτική. Θα ήθελα να πω ότι θα ακολουθήσω στη συζήτηση τη δομή του εγγράφου που έχετε στους φακέλους σας και θα ήθελα να μου μεταφέρετε τις προτάσεις και τις απόψεις σας και αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό σήμερα ευχαρίστως να τις λάβω πριν ακριβώς από την σύνταξη του πρώτου σχεδίου της έκθεσης ώστε να είμαστε όσο πιο δικοδομητικοί γίνεται. Όπως λέγαμε λοιπόν η τεχνολογία έχει επαναστατικές επιπτώσεις στην ζωή μας Προκαλεί δηλαδή πολλές αλλαγές και πολλές μετακινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός αυτής. Κάποιες πολιτικές ήδη υπάρχουν. Κάποιες χώρες μέλη έχουν εντοπίσει την πρόσβαση στην ε, ψηφιακή επικοινωνία ως προτεραιότητα και αυτό αφορά βεβαίως τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και υποψήφιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε πρόσφατα να υπάρχουν και στρατηγικές που αποβλέπουν στην διασφάλιση των ψηφιακών ελευθεριών ως τμήμα της στρατηγικής μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ίδιο αφορά και τα εργαλεία που προσπαθεί να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν σημαντικό να διασφαλίσουμε την ανταπόκριση στις ανησυχίες των πολιτών με τα κατάλληλα εργαλεία. Είδαμε τι έγινε στην κατά την Αραβική Άνοιξη μάλιστα. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τις νέες απειλές ώστε να απολαμβάνουν οι πολίτες ελευθερία μέσω αυτών των τεχνολογιών. Θα πρέπει επίσης να δούμε και θέματα που αφορούν εμπορικές συναλλαγές και ανάπτυξη ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην διπλωματία μας μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών. Θα τονίσω επίσης κάποιες από τις ανησυχίες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε νέες απειλές ασφάλειας. Είδαμε ένα ιό που ονομάζεται flame floga που προέκυψε πρόσφατα. Είδαμε κάτι επίσης σε σχέση με το Ιράν, κάποιες επιθέσεις και θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιος είναι υπόλογος αυτές τις επιθέσεις, ποιοι θα λογοδοτήσουν, σε ποιο πλαίσιο θα γίνει αυτή η προσπάθεια στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ή κάπου αλλού κλπ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης θεωρεί ότι αυτές οι δομές είναι κρίσιμης σημασίας και θα πρέπει να είναι ασφαλείς και διαρκείς. Ταυτόχρονα όμως δεν θα πρέπει να υπερεκτιμήσουμε τις απειλές οι οποίες προέρχονται από αυτές τις νέες μορφές γιατί το επίπεδο φόβου και οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεξέλεκτες καταστάσεις προ την λάθο βεβαίω κατεύθυνση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε προσεκτικά τι γίνεται με την αμέλεια στην παροχή τη απαραίτητη ασφάλεια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει ένα ισοζύγιο, μια ισορροπία μεταξύ ασφάλεια και ελευθερία. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέπουμε ότι η πάλι για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταφέρθηκε στο ίντερνετ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία έκφρασης του λόγου, όπως δημοσιογραφία και όλα αυτά θα πρέπει να ασφαλίζονται και να προστατεύονται. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτό το μεγάλο δυναμικό προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη νέα τεχνολογία, είδαμε ταυτόχρονα να υπάρχουν και προσπάθειες ελέγχου αυτής της έκφρασης μέσω καταστολής, περιορισμού στην ε, ψηφιακή κοινότητα κλπ. κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσπάθειες μέσω των εργαλείων που θα πρέπει να διαθέσουμε στις κοινωνίες μας. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι τα όρια μεταξύ κοινωνιών που αντιμετωπίζουν καταστολή και ελευθέρων κοινωνιών, τα όρια αυτά να συχαίονται. Βλέπουμε ότι έχουμε μεταφορά τεχνολογιών, βλέπουμε να έχουμε διακίνηση ιδεών και βλέπουμε επίσης ότι ότι θεωρούμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ότι λείπει διαφάνεια σε αυτές τις κοινωνίες που αντιμετωπίζουν αντικαταστολή, ότι λείπει διαφάνεια και λογοδοσία και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει με αυτά τα εργαλεία που αντιμετωπίζουμε, που αναπτύσσουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Εμείς λοιπόν ως δημιουργοί πολιτικής δεν μπορούμε να δράσουμε μόνοι μας, γιατί όλες οι υποδομές, το hardware, το software, οτιδήποτε αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτρέπει τη σωστή επαφή και συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μεταξύ κοινωνίας των πολιτών και χρηστών των ψηφιακών μέσων. Θα πρέπει επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερες προσπάθειες για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Είχαμε πρόσφατα το παράδειγμα της ε, Vodafone που υποχρεώθηκε από το καθεστώς Μουμπάρακ ε, να περιορίσει το δίκτυο ώστε να καταστήλει την εξέγερση. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα προλάβουμε και να τα αντιμετωπίζουμε. Εκτός λοιπόν από τις δικές μας πολιτικές έχουμε και την αυξανόμενη πρόκληση της, διακυβε... της κυβερνητικής διακυβέρνησης. Δηλαδή το πώς θα πρέπει να διασφαλίσουμε αφενός το να μείνει ανοιχτό το ίντερνετ και να λειτουργεί και αφετέρου να το προστατεύσουμε από απόπειρε που προέρχονται από αναπτυσσόμενες δυνάμεις παγκοσμίω που αποβλέπουν και αποσκοπούν στον έλεγχο του ίντερνετ. Είναι λοιπόν σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική και ξεκάθαρη ιδέα για το θα πρέπει να κάνουμε εκεί ώστε να συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκόμενους και να έχουμε μια προσέγγιση σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, με τις επιχειρήσεις, με τους χρήστες ώστε ακριβώς να αποτρέψουμε τη χειραγώγηση του διαδικτύου και τις απόπειρες κατά της ε, κυβερνητικής διακυβέρνησης, διακυβέρνησης του κυβερνοχώρου. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για τις εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αντίκτυπο που έχει όλο αυτό το ζήτημα εκεί. Μίλησαμε σήμερα για ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε πολιτικές οι οποίες θα είναι αξιόπιστες παγκοσμίω. Δεν μπορούμε λοιπόν να διαχωρίζουμε εσωτερικές με εξωτερικές πολιτικές. Θα αναφερθώ σε δύο τομείς που παρουσιάζουν μεγάλες ευκαιρίες και μετά θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις και για την ανάπτυξη στις στοχές χώρες του κόσμου οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες. Μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κρίσεις, ανθρωπιστικές κρίσεις ή σε θεομηνίες μέσω των νέων τεχνολογιών που θα μας βοηθήσει στην αντιμετώπιση τους. Επίσης θα πρέπει να καλύψουμε το ψηφιακό χάσμα. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες να έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή κοινότητα ώστε να έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση, σε υγεία, να βρουν δηλαδή, τους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάστασή τους. Για την παρουσία μας τώρα στην ως Ευρωπαϊκή Ένωση στον υπόλοιπο κόσμο, νομίζω θα πρέπει να δούμε εδώ πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες στην διπλωματία. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ώστε να καταπολεμήσουμε τον εξτρεμισμό, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διάφορα εργαλεία όπως το Ευρωπαίανα, το οποίο είναι μια ιστοσελίδα που περιλαμβάνει πολιτιστικό περιεχόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα μπορούσε να βοηθήσει όταν κάνουμε δράσεις ή όταν σχεδιάζουμε δράσεις εξωτερικές. Το ίδιο ισχύει επίση και για τι ευκαιρίε που έχουμε εμεί εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα όγκο πληροφοριών που βρίσκεται στα θεσμικά όργανα εδώ τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούμε να μοιραστούμε και το οποίο είναι σημαντικό και για αυτού εντό αλλά και για αυτού εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω τη χρήση νέων τεχνολογιών που θα επιτρέπει την χρήση ανοιχτών στοιχείων, ανοιχτών δεδομένων που αποδεικνύει την διαφάνειά μα. Δηλαδή καλούμε τον κόσμο να σχολιάσει τη δουλειά μα και αυτό βεβαίω δεν περιορίζεται στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλήγοντας λοιπόν νομίζω θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τις πολιτικές μας ώστε να δώσουμε τη δύναμη που χρειάζονται οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να γίνουν όλα αυτά με έναν τρόπο στρατηγικό με τη συμμετοχή των πολιτικών, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και βεβαίως προσβλέπω στην συνεργασία μαζί για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Υπάρχει ένα παράδοξο ε, στο να παρακολουθούμε την τεχνολογία που όμως μας προσφέρετε εσείς. Όσο πιο προηγμένη τηλεφωνία, τόσο πιο πολύ και ο έλεγχος, τον οποίο ε, υφιστάμεθα, αλλά εν Η κυρία Λάτφορτ. Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική έκθεση πιστεύω και συγχαίρω τη συνάδελφο για τη δουλειά της. Στο έργο Για το θέμα αυτό, το οποίο είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα όμω να κάνω δύο σχόλια. Στη σελίδα 3 η αναφορά στο Flame και το Stuxnet. που πιστεύουμε ότι αφορά περισσότερο διαρροές από το λευκό οίκο. Τουλάχιστον αυτό λένε οι New York Times και δεν έχουν διαψευστεί. Ούτε έχουν επιβεβαιωθεί βεβαίω. Ίσως λοιπόν οι Ηνωμένε Πολιτείε μαζί με το Ισραήλ, ίσως μαζί με το Ισραήλ, όχι μόνο ανέπτυξαν, αλλά χρησιμοποίησαν το στάξινε τη βάρο του πυρηνικού προγράμματο του Ιράν. Στάξτε το οποίο θεωρείται, ε, μάλλον το Ιράν το οποίο θεωρείται ότι είναι υπεύθυνο για το Φλέιμ. Και χωρίς να είμαι ειδική στα τεχνικά, στη νέα τεχνολογία, το Φλέιμ έχει σαν συνέπεια ή σαν σημασία ότι μπορούν να μπουν ή ε, και ε, μέσα σε ένα σύστημα και το ε, σύστημα αντιβάρους, το αντιϊκό, να μην τους συλλάβει. Αυτό είχε συμβεί ήδη πριν από κάνα δύο χρόνια. Και διέλαθε των ε, εφιών αυτών τεχνοκρατών η εισαγωγή ιών αλλά επίσης θα ήθελα να αναφερθώ και στην διάσκεψη που είχαμε με, την, με το κυβέρνο έγκλημα. Με τον ειδικό κυβερνό εγκληματολόγο της κυρίας Άστον, του οποίου το όνομα δεν τολμώ να προφέρω γιατί είναι αισθονός. ο οποίος είχε αναπτύξει την κυβερνοάμυνα στην Εστονία και μετά στο ΝΑΤΟ και τώρα στην κυρία Άρστον. Φαίνεται ότι είναι πολύ δυνατός. Και κατά τη συζήτηση εκείνη μας είπαν ότι υπήρχε μια τριημερής ε, ε, στο ΝΑΤΟ με ύψιστου επίπεδου ειδικού και νομικού δικηγόρου για το κατά πόσον το κυβερνοέγκλημα, ακριβώ αυτό το θέμα, α, συνιστά πράξη πολέμου. Μου είχαν υποσχεθεί και κάτι links, αλλά δεν τα έλαβα ακόμα. Πριν από δύο εβδομάδε έγινε αυτή η συζήτηση. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι με το να δίνονται διαφορετικές τοποθετήσεις, δηλώσεις, βεβαίωσεις, είναι σαν να αλλάζουμε διαρκώ τους κανόνε του παιχνιδιού. Άρα μπορεί να έχουν αναπτύξει οι ΗΠΑ ε, κυβερνό όπλα, αλλά το θέμα είναι να τα έχουν αξιοποιήσει κιόλα. Εκεί είναι το ζήτημα. Και εκεί βέβαια γίνεται και η σύγχυση για το πώ μπορούμε τον κυβερνό πόλεμο να τον αντιμετωπίσουμε. Πότε χαρακτηρίζεται πράξη πολέμου, ένα κυβερνό έγκλημα, πώς θεωρείτε ότι έχουν εμπλακεί και από πότε αρχίζει να εφαρμόζεται το ποινικό δίκαιο εις βάρος μιας χώρας. Και χωρίς να είμαι ειδική, παρακολούθησα λίγο αυτόν τον διάλογο, τον διατλαντικό για το, υπερ... για το αλλά πώς θα αντιμετωπίσουμε τις κυβερνοεπιθέσεις εις βάρος ημών όταν οι Δύση, οι αναπτύσσουν κυβερνοεπιθέσεις προς άλλους. Δεν έχω απαντήσεις φυσικά. Αλλά αν η συνάδελφος δεν ε, είχε υπόψη σε αυτή τη διάσκεψη, ας την ε, κοιτάξει. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μας απασχολήσει το τι θα πράξουμε περαιτέρω. Ξέρουμε ότι οι Ρώσοι και οι Κινέζοι μπορεί να έχουν ε, προσχωρεί στη Εθνή Σύμβαση για το Κυβερνοέγκλημα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση τους υποψιάζεται ότι προσπαθούν με τον τρόπο αυτόν να αποκρύψουν στοιχεία και την ε, δυνατότητα την οποία επιδιώκουν ε, για απεριοριστή πρόσβαση στο ίντερνετ. Μάλλον να περιορίσουν για, για τους πολίτες τους την πρόσβαση στο ίντερνετ. Πώ λοιπόν εμεί θα πείσουμε του εχθρού μα ή θα αντιμετωπίσουμε του εχθρού μα όταν οι φίλοι μα είναι αυτοί που διαπράττουν αυτά τα κυβερνοεγκλήματα. εγκλήματα. Επίσης στην τεχνολογία απλής χρήσης, γιατί είχαμε και τη δυτή χρήση νωρίτερα και της, ε, της πολεμικής δηλαδή και μη χρήσης τεχνολογία και τις άδειες ε, για την ε, εμπορία αυτών των προϊόντων. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε τεχνολογία ε, εξαιρετικά προηγμένη, εξαιρετικά επικίνδυνη, που εξάγεται βέβαια. Ασφαλώς τη διαθέτουν ή την αποκτούν και οι δικές μας μυστικέ υπηρεσίε, Αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε να κυκλοφορεί ε, ένα σύνολο, ένα οπλοστάσιο τόσο επικίνδυνο σε ε, απλούες εμπορικές εκθέσεις ανά την Ευρώπη. Δεν θα έπρεπε να ελέγξουμε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούν τα προϊόντα αυτά και δεν θα έπρεπε να ελέγξουμε κάπως και τις τηλεπικοινωνίες στο επίπεδο αυτό. Προτάσεις μόνο. Κύριος Πάσκου. Εν γέννη, όποιος θέλει να έχει αποτελεσματική παρακολούθηση, καλό θα είναι να αφήνει τον κόσμο να εκφράσει όσο δυνατόν πιο ελεύθερα. Η κυρία Οιούλαντ. Πρόεδρε, ενδιαφέρουσα η έκθεση. Πολλά θα ήθελα να πω, που τα κάλεψε όμως η Σάρα για την κυβερνοασφάλεια ιδιαίτερως. η οποία πιστεύω αξίζει και χρειάζεται μια χωριστή έκθεση. Υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα στην έκθεση αυτή που θα μπορούσαν να εξεταστούν αυτόνομα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται οπωσδήποτε να εργαστεί υπερστορές βάθος, πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εστιασμένα στην κυβερνό ε, ασφάλεια, διότι οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται μέρα με τη μέρα. Αν παραμείνει λοιπόν το τμήμα αυτό στην έκθεση, στο πρώτο στάδιο, θα ήταν καλό ίσως να δούμε και το τι πράττουν άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμοί, τι είδους έρευνα, τι είδους τεκμηρίωση έχουν, θα αναφερόμουν παραδείγματι στο κέντρο της για την κυβερνοασφάλεια στο Ταλήν της Εστονίας που συνεργάζεται με τον ΝΑΤΟ εδώ και πολύ καιρό για τα θέματα αυτά και ιδιαιτέρως μελετά εφιστάμενη νομοθεσία και συγκρίνει η νομοθεσία που ισχύει μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό θα ήταν χρήσιμο, αλλά και άλλοι οργανισμοί. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Και επίσης, όταν μιλούμε για κυβερνοασφάλεια, θα πρέπει να καλούμε και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεργάζονται στενότερα στον τομέα αυτών. Γιατί ναι, είναι μια κοινή απειλή, το ξέρουμε αυτό όλοι. Αλλά ταυτόχρονα Ίσως θα ήταν και ένας τρόπος να επιτευχθεί περισσότερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών. Ένα άλλο ζήτημα που είναι η αξιοπιστία για μένα, πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, όταν μιλούμε για κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για ελευθερίες που αναφέρατε κι εσείς πολλές φορές. Θα πρέπει κι εμείς ιδιαίτερως να προσέχουμε για το πόσο μπορούν, μέχρι ποιου βαθμού μπορούν να καταγράφουν, να παρακολουθούν ε, τηλεπικοινωνίες και κίνηση στο διαδίκτυο οι μυστικέ υπηρεσίες. Αυτό θα θέμα έχει απασχολήσει πολύ την κοινή γνώμη στη χώρα μου. Ήδη ο Πρωθυπουργό το έθεσε. Το πόσο ελεύθεροι είμαστε και πόσο ασφαλείς. Γιατί εάν δούμε την ελευθερία στο διαδίκτυο ως ανθρώπινο δικαίωμα, και την προβάλλουμε και μέσα από την εξωτερική μας πολιτική, την κοινή εξωτερική πολιτική, προσπαθώντας να παρουσιάσουμε ένα θετικό πρότυπο για τις λοιπές χώρες ανά τον κόσμο, πριν το πράξουμε αυτό, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε τακτοποιήσει τα του οίκου μας. Και αυτή είναι και μια άλλη πτυχή. Ένας άλλος τρόπος να δούμε το τι θα μπορούσαμε από, ε, χωριστά ίσως να δούμε ε, Ω ως συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής μας και των άλλων σχετικών ε, επιτροπών. Προστασία δηλαδή των ανθρωπινών δικαιωμάτων για τους πολίτες μας. κυρία Γκόμες έχει το λόγο. I, I think it's very Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες της Μαρία για την ψηφιακή ελευθερία πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν θα έχουμε ψηφιακή ελευθερία χωρίς ασφάλεια. Είναι μια βασική ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί. Στη νέα τάξη ειδικά την οποία, στην οποία βρισκόμαστε και όπου εξαρτώμαστε όλο και περισσότερο από την τεχνολογία. Τίποτα δεν γίνεται τώρα χωρίς τον κυβερνοχώρο. Παρά τις απόπειρες διαφόρων κρατών να περιστήλουν τις ελευθερίες ε, στον κυβερνοχώρο, με απειλή της ανθρώπινης ελευθερίας, παρόλα αυτά υπάρχει μια πολυμορφία μη κρατικών φορέων που υπάρχουν στον κυβερνοχώρο, που κανένας δεν τους ελέγχει και που αυτοί για διάφορους λόγους μπορεί να επιδιώξουν να περιστύλουν την ε, ελευθερία μας, ε, ακόμα και το δικαίωμα στη ζωή, ε, χειραγωγώντας, χρησιμοποιώντας με διαφόρους τρόπους το κυβερνοχώρο. Ήμουν σε μια συνάντηση με εμπειρογνώμονες που, μίλησαν, μιλούσαν για τη δημιουργία στην Europol ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταπολέμησης του Κυβερνοεγκλήματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα δοθούν τα χρήματα από τα κράτη-μέλη για να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο, γιατί χρειάζονται χρήματα. Και πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε και τα κράτη-μέλη, ε, γιατί υπάρχει πραγματικά ανάγκη να συνεργαστούν για, και να γίνουν αποτελεσματικά με σεβασμό των βασικών ελευθεριών από τη μία, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε άλλους να απειλήσουν αυτές τις ελευθερίες. Μιλάμε για κυβερνοεγκλήματα που αφορούν την εκμετάλλευση παιδιών για σεξουαλικούς λόγους. The safety of our nuclear Που απειλούν ακόμα και τις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις και την ασφαλειά τους. Και εκεί πέρα, σε αυτό το ε, φάσμα, ε, μπορούν να μπουν τα πάντα. Το πώς λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ε, οτιδήποτε. Όπως είπε και η Σάρα, στη συναντήση με τους Αμερικανούς ομολόγους μας, συνειδητοποιούμε πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Παρότι μπορούμε να συνεργαστούμε και πρέπει να συνεργαστούμε σε πολλά πράγματα και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτή τη συνεργασία, βλέπουμε τις διαφορές. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν τα όρια που πρέπει να υπάρχουν ανάμεσα στις βασικές ελευθερίες και στην προστασία της ιδιωτικής σφαίρας από τη μία και την ασφάλεια στην άλλη. Αλλά υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Και εμείς πρέπει να καταλάβουμε τι διακυβεύεται εδώ. Τι διακυβεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Φυσικά οι εμπειρίε όλων μα δεν είναι οι ίδιε. Δεν έχουμε εμεί τι εμπειρίε που είχαν οι Εσθονοί, αλλά οι δυνατότητε να ε, παρισφρήσουν ε, στη ζωή μα, στην ποιότητα τη ζωή μα κυβερνοεγκληματίε είναι αισθητοί. Οι αισθητέ. Επίσης, ακόμα και ε, στην εξωτερική πολιτική μπορούν να παρέμβουν, γιατί ζούμε σε ένα ε, παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Μάλιστα. Α, πρέπει να δούμε ποια είναι αυτή η ισορροπία λοιπόν ανάμεσα στην ε, ασφάλεια και στις ελευθερίες. Ο κ. Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συγχαρώ την ησυχήτρια για αυτή την προκατακτική δουλειά πριν από την παρουσίαση της έκθεσης. Νομίζω ότι Πρόκειται για μια έκθεση για ένα νέο θέμα που μας αφορά και παρουσιάζεται σε ένα έγγραφο καλά δομημένο που καθορίζει συσχετισμούς με σημαντικά άλλα θέματα και θέτει και κάποια λειτουργικά ζητήματα. Νομίζω ότι οι παράμετροι του ίντερνετ έχουν αλλάξει τελείως την καθημερινή μας ζωή και εδώ εξετάζουμε θέματα που αφορούν βεβαίως την ασφάλεια και την ψηφιακή ελευθερία. Στο πλαίσιο αυτό η κυρία νομίζω σωστά έδωσε έμφαση στην ε, σημασία που έχει αυτή η νέα πραγματικότητα. Έχουμε δηλαδή στρατούς που δεν αντιμετωπίζουν ορατούς εχθρούς και έχουμε και εχθρούς που δεν έχουν στρατό. Τα κυβερνοεγκλήματα λοιπόν, οι κυβερνοεπιθέσεις είναι σωστά παραδείγματα και η Εστονία είναι το πιο δεκτικό. Άλλα θέματα που εξετάζουμε το πρόβλημα είναι το θέμα τη ψηφιακή ελευθερία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάμε πραγματικά για την Αίγυπτο, την Κίνα, την Συρία, την Τινησία. Θέματα που αφορούν βέβαια άμεσα την Αραβική Άνοιξη. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να συμπληρώσουμε αυτέ τι αναφορέ στα ανθρώπινα δικαιώματα με μια μελέτη που έκανε το ΙΡΙ με 786 ενήλικε στην Κούβα, σε διάφορες επαρχίες της ε, χώρα αυτής, όπου ρωτούσαν αυτούς του κουβανού πολίτες σε σχέση με δυνατότητα πρόσβασης ε, στο ίντερνετ και στην κινητή τηλεφωνία. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η εμπειρία αυτή και να, θα πρέπει να την περιλάβουμε. Εξετάζουμε επίσης το θέμα της ε, διακυβέρνηση του κυβερνοχώρου. Εδώ εμπλέκονται διάφοροι παράγοντες θέμα που αφορά και τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί ξέρουμε ότι πάρα πολλέ μεγάλε επιχειρήσει έχουν έδρα τι Ηνωμένε Πολιτείε, όπου έχουμε συχνά θέμα δικαιοδοσία. Όμω, ημερίζομαι τον στόχο μα θέτει η συγκήτρια, από την έννοια δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει ένα ηγετικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει και ένα ζήτημα κλειδί που αφορά το εμπόριο και τι εξαγωγέ. Μιλάει για μόνιμες, μόνιμους περιορισμούς όσον αφορά κάποια εμπορικά προϊόντα και για τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Νομίζω θα πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στις νόμιμες θέσεις με τις καθαρά νομικές δυνατότητες. Εδώ νομίζω ότι επιβάλλεται η ανάγκη καθορισμού κανονών παιχνιδιού που θα πρέπει να είναι σαφείς και ξεκάθαρη και που θα ακολουθούν κατευθείαν γραμμές από την Κομισιόν. Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει κυρώσεις εμπορικές. Εδώ έχουμε λοιπόν στα πλαίσια της κρίσης ανάγκη για κανόνες ξεκάθαρους και όπου θα πρέπει να συμμεριζόμαστε και να συνδέουμε την ηθική με τους κανόνες. Νομίζω είναι ενδιαφέρον επίση το θέμα τη ψηφιακή διπλωματία, παρόλο που νομίζω ότι αυτό το εργαλείο είναι κάτι το οποίο προσανατολίζεται περισσότερο και αφορά περισσότερο τα θέματα τα πολιτιστικά. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι ανοίγει μια ενδιαφέρουσα δυνατότητα επικοινωνίας που ήδη κάποιοι βουλευτές χρησιμοποιούμε ας πούμε στα πλαίσια της Eurolat, της κοινοβουλευτικής διάσκεψης, τα μέσα, τα ψηφιακά μας επιτρέπουν να προχωράμε. Και ίσως αυτό το κεφάλαιο της ψηφιακής διπλωματίας πέρα από την πολιτιστική διάσταση θα μπορούσε να συνεισφέρει με κάποια πολύ σημαντικά εργαλεία όπως ακριβώς αυτό μας προτείνει η συγγήτρια. Τέλος, σχετικά με την γενική αρχή να μην περιορίζουμε ενδεχομένως τις τεχνολογίες οι οποίες είναι υπέρ της ελευθερίας τότε βεβαίω αυτό θα πρέπει να το εντάξουμε σε ένα συγκεκριμένο εμπορικό πλαίσιο. Μιλάμε για συμφωνίες συνεργασίας ή συμφωνίες σύνδεσης με σημαντικό εμπορικό περιεχόμενο. Βεβαίω αυτό η γενική αρχή είναι σωστή, αλλά βεβαίω να την θέτουμε στο σωστό πλαίσιο συμφωνία δηλαδή ΕΕ με τρίτε χώρες. Τέλος Πρόεδρε, να καταλήξω λέγοντας ότι ζούμε την ε, τεχνολογική εποχή, την εποχή την ε, πυρηνική, την εποχή του ίντερνετ. Όμως όλη αυτή η τεχνολογική πρόοδος δεν κατάφερε να αλλάξει τη συνείδηση και τη φύση του ανθρώπου που δεν οδηγεί στην βελτίωση του κόσμου. Κόσμος που συνδέεται και με το κόσμιος. Δεν έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτό το σημείο. Οπότε, Πρόεδρε, νομίζω οι διαστάσει που αναφέρει η συγγήτρια είναι σωστέ, τι συμμερίζομαι και βεβαίω συμμεριζόμαστε όλοι την ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ένα ηγετικό ρόλο σε αυτό το τομέα που είναι τόσο σημαντικό και τόσο καινοτόμο. Οπότε πρέπει να αναπτύξουμε και σωστέ πολιτικέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το πρόβλημα είναι, ασφαλώ το ξέρετε, ότι οι νέοι όλο και μαζεύονται για να μπορούν να κάτσουν μαζί και να παίξει ο καθένα με το παιχνίδι του, το ηλεκτρονικό, και έτσι διερωτώμεθα γιατί μαζεύονται και συναντιούνται. Αλλά μπας περιπτώσει, κυρία Σάκε. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις αρχικές ε, παρατηρήσεις. Ένα πράγμα νομίζω καθίσατε σαφές και θα ήθελα να το διευκρινίσω προκαταβολικά γιατί του παρατηρήσει αφορούν το θέμα της ασφάλειας. Ε, ανέφερε και ο Πρόεδρος ήδη ότι υπάρχει άλλη έκθεση σε επίπεδο Επιτροπής Άμυνας ε, για την ασφάλεια. Και άρα όλο τον όγκο των θεμάτων ε, στις λεπτομέρειές τους τον αφήνω για την έκθεση ΣΕΔΕ αλλά φυσικά δεν μπορώ και να αποκλείσω από τη συζήτηση, γι' αυτό έχω αυτή την σύντομη αναφορά στο θέμα της ασφάλειας. Για την κυρία Γκόμες αυτό που μας διδάσκει η προσέγγιση ως προς τον ε, πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, επί παραδείγματι, είναι ότι κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη για λήψη μέτρων ε, αποτελεσματικών, αλλά διαπιστώνεται ότι το να περιστέλουμε τις ελευθερίες μας εν τέλει αποβαίνει αντιπαραγωγικό και εσφαλμένο και μάλλον βοηθά τους εχθρούς μας παρέμας. Αυτό και για την ε, κυρία Λάτφορτ και την παρατήρησή της τη σχετική με τους Ιού, την προέλευσή τους και τον τρόπο με τον οποίο η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να του αντιμετωπίσει. Ναι, για τη διάσκεψη ναι την παρακολουθώ. Θα πρέπει να δούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς ε, εστιάζει στα θέματα αυτά και πώς ε, αντιμετωπίζει τα προβλήματα και αυτό όχι μόνο σε επίπεδο μελών αλλά και, και κυβερνήσεων αλλά και ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων κτλ. και για την κυρία Όιλαντ και την ερώτηση της, ε, σχετική με την αξιοπιστία. Νομίζω ε, είναι η απάντηση ίδια. Κύριε Σελαφράνκα, νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για, περισσότερα, για περισσότερη πρόοδο στον τομέα της διπλωματίας. Συμφωνώ επίσης μαζί ότι η τεχνολογία έχει αλλάξει τη ζωή μας, χωρίς όμως να αλλάξει την πεμπτουσία της ανθρώπινης φύσης. Και γι' αυτό όταν αντιμετωπίσουμε μια νέα μια κατάσταση θα πρέπει να δούμε αν είναι τελείως καινούρια ή αν απλώς εφαρμόζονται κατά διαφορετικό τρόπο νόμοι και πολιτικές επειδή έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα. Το ίδιο και για την κυβερνοασφάλεια. Υπάρχουν εγκλήματα τα οποία διαπράττονται μέσω του ίντερνετ. Χρησιμοποιούν ω μέσο το ίντερνετ. Παραδείγματι, η πώληση online προϊόντων ε, Εγκλήματο, κλοπημαίων φερπίν. Αλλά δεν είναι το ίδιο αυτό με το έγκλημα, το οποίο διαπράτεται μέσω του ίντερνετ. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο προσεκτική και να μην απομακρυνθώ από τι ευρωπαϊκέ αξίε στην ε, παρουσίαση του σχεδίου. Αυτό είναι τα τελευταία μου σχόλια σχέση με τι ε, εξαγωγέ αυτέ σε περίοδο κρίσεω, ε, γιατί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ούτω ή άλλω δεν είναι καλό πράγμα η υπερβολική επιβολή κανόνων και διατάξεων, ούτε για τον πολίτη, ούτε για τις επιχειρήσεις, ούτε τελικά για τον τρίτο αποδέκτη. Το γραφειοκρατικό βάρος και η υπερβολική, υπερβολικά περίπλοκες διαδικασίες δεν ε, είναι μια καλή λύση. Μάλλον θα πρέπει να τους αποφύγουμε. Ταυτόχρονα, στα όσα είπε και η κυρία Λάτφορτ για, τα, για τις τεχνολογίες απλής ή διπλής χρήσης, ε, ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμεθα το θέμα αυτό νομίζω δείχνει και το τι είδους Ευρώπη είμαστε. Ποια Ευρώπη είμαστε. Και δεν θέλω να το εξηγήσω λίγο περισσότερο. Το χάσμα δηλαδή μεταξύ των αρχών μας και της πρακτικής μετατρέπεται και σε κυρώσεις αλλά και στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε ζητήματα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε αντίστοιχη ζημιά. Άρα πρέπει να πάνω πρώτα να ψωθήσουμε να είμαστε αξιόπιστοι, να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας και να αποφύγουμε να ενισχύσουμε τους εχθρούς μας, ώστε αυτοί να καταπιέσουν τους ίδιους πολίτες ή να προσβάλλουν περισσότερο τις δραστηριότητες των δικών μας επιχειρήσεων ε, μέσω μαζικής ε, παρακολούθησης και ε, ως εκ τούτου νομίζω ότι είναι ένα μέτρο δύσκολο, αλλά μπορούμε να βρούμε τις λύσεις με καλά στοχευμένες πολιτικές. Θα προσπαθήσω να το διατυπώσω όλα αυτά στο σχέδιό μου. Πολύ σύντομα θα σας το καταθέσω. Μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού έχω προθεσμία. έχουμε προθεσμία για τις τροπολογίες 29 Αυγούστου για να ψηφίσουμε τον Σεπτέμβριο σε εύχομαι να περάσετε καλό καλοκαίρι φυσικά, αλλά θα χρειαστεί να αφιερώσετε και λίγο χρόνο στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ. Πριν ε, σταματήσουμε, θα ξαναρχίσουμε τη συνεδρίασή μας ε, στι 3. Τρία θέματα έχουμε, την κατάσταση στη Συρία, στην Αίγυπτο και στο Μπαχρέιν. Αυτά τα ξαναλέμε στις 3.